Καθίστε παρακαλώ. Ο κύριος Κράμερ, ως άλλος για Ζεμπόφσκι από το παρελθόν, επιμένει να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας το ταχύτερο δυνατό. Άφησα βέβαια δύο λεφτά τζόγο, γιατί κάποια μέλη έχουν ακόμα δυσκολίες για να φτάσουν μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα το πρωί. προβλήματα κυκλοφορίας στην πόλη των Βρυξελών. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω τι ανακοινώσει του Προέδρου. Και να σας πω καταρχήν ποια είναι τα συμπεράσματα που προήλθαν από τη συνεδρία στο συντονιστό χθε το βράδυ. για τους εισηγητές καταρχήν, το διορισμό των εισηγητών. Είχαμε τρεις εκθέσεις και οι τρεις μη νομοθετικού περιεχομένου. Και εδώ η σύσταση των συντονιστών είναι να μην καταρτήσουμε καμία έκθεση για τα θέματα αυτά, επομένως δεν λαμβάνουμε καμία δράση. Πρόκειται για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων, είναι μια, το ένα θέμα η μοναδικότητα των διπλωμάτων οδήγησης και επίσης το έγγραφο της Κομισιόν για τα δεδομένα για, τα, για τις θαλάσσιες μεταφορές και τέλος το έγγραφο εργασίας της Κομισιόν για το ασφαλές εμπόριο και την ηλεκτρονική σάρωση των κοντέινερς. Θεωρείται ότι αυτό είναι ένα καθαρά στατιστικού χαρακτήρα έγγραφο και δεν χρειάζεται καμία συνέχεια από τη δική μας πλευρά. Εάν δεν έχετε πρόβλημα λοιπόν μπορώ να περάσω στο επόμενο θέμα. είχαμε μία συζήτηση μεταξύ των συντονιστών για τα προφορικά ερωτήματα και συγκεκριμένα το προφορικό ερώτημα για την μαύρη λίστα αερομεταφορέων. Η άποψη των συντονιστών θα ήταν ότι μετά τα τελευταία γεγονότα θα πρέπει να προβλέπουμε και μία προφορική ερώτηση για την εφαρμογή του συνδυοδομικού πακέτου ή των πακέτων και εκεί θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα όχι ότι θα ξεχάσουμε τη μαύρη λίστα των αερομεταφορέων, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε να φέρουμε στην Ολομέλεια του Μαρτίου μια προφορική ερώτηση για τα συνδρομικά πακέτα και μετά η ερώτηση για τη μαύρη λίστα να πάει αργότερα αν θέλει ο Θεός την μήνυ Ολομέλεια του Μαρτίου ή την Ολομέλεια του Απριλίου για την μαύρη λίστα στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Αυτή είναι λοιπόν η πρόταση των συντονιστών. Ομόφωνη άποψη όλων των συντονιστών. Εάν συμφωνείτε λοιπόν θα πράξουμε ούτω. Κύριε Κούν, έχετε να πείτε κάτι. Μονάχα για τα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε. Και το είχα αναφέρει στη συζήτηση ότι η πρόταση του ΕΛΚ και αυτά που είχε ζητήσει ο κύριος Ντεβεράκ δεν είχαν τύχη ανταπόκριση, αλλά τελικά εμεί συμφωνήσαμε με την τελική πρόταση. Απλώ θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά ότι δεν έτυχαν ανταπόκριση στι προτάσει του κύριου Ντεβεράκ. Ευχαριστώ. Αυτό αφορούσε κάποιο στοιχείο του κειμένου το οποίο εμεί είχαμε προτείνει. Και να σας πω επίσης ότι προσεκλήθησαν οι συντονιστές να υποβάλουν προτάσεις για την προφορική ερώτηση για το συνδυοδομικό πακέτο μέχρι, μέχρι την Τετάρτη. Ώστε να προσπαθήσουμε να το ετοιμάσουμε. Σε εσά εναπόκειται λοιπόν από τις πολιτικές σα ομάδε να κάνετε τι απαραίτητε συνεννοήσεις. Το άλλο θέμα που εξετάστηκε ήταν η προετοιμασία του, των κατευθυντήριων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Είχα ζητήσει από τους να έχουμε τακτικές απόψεις για το θέμα αυτό. για τη μεταρρύθμιση των κατευθυντήριων γραμμών, ώστε να προετοιμαστούμε για την στιγμή που θα είχαμε τις ε, προτάσεις της Κομισιόν για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Η ιδέα είναι να παραμείνουμε ενήμεροι με τα τεκτενόμενα στον τομέα αυτό και συμφώνησαν οι συντονιστές να ακολουθήσουμε αυτή την, ε, αυτή την ε, πορεία. Ένα καφέ παρακαλώ. Ναι, Μιχάλη, συγγνώμη. Θα ήθελα να υπενθυμίσω για μια ακόμα φορά ότι δεν υπήρξε κάποια μεγάλη αλλαγή. Αυτά τα οποία είχα πει για το Transrapid ισχύουν, αλλά επίση και ο διάδρομο Παλέρμο-Βερολίνο θα πρέπει να επεκταθεί μέχρι και την Στοκχόλμη. Τα είχα πει αυτά χθε, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι χρήσιμο να το έχουμε στο μυαλό μα άμα γίνει η αναθεώρηση των κανόνων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ευχαριστώ, Μάικελ. Εγώ νομίζω ότι όταν γίνει η μεταρρύθμιση τα πάντα παίζονται. Επομένω, ο κάθε βουλευτή έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του όπω έχει κάνει εσύ στο παρελθόν ήδη για αυτά τα σχέδια. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι όμως όταν έρθει η Κομισιόν με τις προτάσεις της, αντί να περιμένουμε να έρθουν αυτά για να αντιδράσουμε, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι αμέσως να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας. Για τα προγράμματα της ΣΤΟΑΣ προτάθηκε ο κύριος Κόκ και η κυρία Τικαού να είναι οι εκπρόσωποι μας και ζήτησα να συνεννοηθούν με τους συντονιστές για να θέσουν προτάσεις και τροποποίηση των προτάσεων που βρίσκονται στο φάκελό μας σε σχέση με την ΣΤΟΑ. Έτσι οι πολιτικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν προτάσεις. Έχουμε λοιπόν τώρα, όπως είπα, την κυρία Τικάου και τον κύριο Κόκ που είναι οι εκπρόσωποι μας στην ΣΤΟΑ, στο πάνελ της ΣΤΟΑΣ όπου μπορούμε να επηρεάσουμε τις μελέτες οι οποίες θα, θα καταρτιστούν. Επίσης, έχουμε λάβει μία αναφορά για την οδική ασφάλεια στην Ιρλανδία μέσω της Επιτροπής Αναφορών. Αυτό δημιουργεί ένα μικρό προβληματάκι, γιατί είναι μία αναφορά που πρέπει να τη λάβουμε στα σοβαρά όταν διαβιβάζεται σε εμά. Αλλά είναι ένα ιδιαίτερα τοπικό θέμα, ενοριακό σχεδόν θέμα θα έλεγα, στην Ιρλανδία σε σχέση με την οδική ασφάλεια. Αυτό το οποίο προτείνουν οι συντονιστέ να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε μεν την αναφορά αυτή, αλλά μέσα στα πλαίσια μιας έκθεσης ιδίας πρωτοβουλία για το πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια, που θα το εγκρίνει η Κομισιόν περίπου τον Ιούνιο του 2010, ώστε <clears throat> επί τη βάση αυτή να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το θέμα αυτό στην έκθεση πρωτοβουλία μα και να συμπεριλάβουμε και το περιεχόμενο αυτή τη αναφορά που αναφέρεται στην Ιρλανδία. Φοβάμαι ότι αν αρχίσουμε να εξετάζουμε συγκεκριμένε αναφορέ από μικρέ γεωγραφικέ περιοχέ για θέματα όπω είναι η οδική ασφάλεια, μπορούμε να περάσουμε τα πέντε χρόνια τη θητεία κοιτάζοντα κάθε ρήμην και κάθε αγιάν τα περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από λοιπόν στην Επιτροπή Αναφορών θα εξετάσουμε το θέμα αυτό σαν τμήμα τη εκθέση πρωτοβουλία μα για το πρόγραμμα οδική ασφάλεια. Αυτή ήταν η απόψη των συντονιστών. Σύμφωνοι. Επιτροπολογία. Οι δύο μόνιμοι εισηγητέ μα θα κοιτάξουν τα στοιχεία που πήραμε από την Διεθνή Ένωση για τι οδικέ μεταφορέ και για τι κατεχώρηση πράξη από την ε, συνθήκη τη Λισαβόνα. Θα έρθουν οι συντονιστέ μα πάλι σε επαφή με τον κύριο Σάγερ, ο οποίο είναι ο εισηγητή τη Νομική Επιτροπή και ο οποίο έχει πάρει την εντολή από τη Συνέλευση των Προέδρων να δίδει <clears throat> κατευθυντήρε γραμμέ για αυτέ τι κατεχώρησει πράξει. Περιμένουμε την ε, πρόταση του κυρίου Σάγερ για αυτό που παλιά λέγονταν επιτροπολογία και τώρα λέγονται κατεχώρηση πράξη. Ο Κράμερ. Τι θα κάνουμε τώρα με τα υγρά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το θέμα αυτό βρισκόταν στην παλιά επιτροπολογία, διαδικασία επιτροπολογίας. Δεν υπήρχε η συνθήκη της Λισαβόνα όταν εξετάσαμε το θέμα των υγρών. Τώρα όμω έχουμε μια νέα διαδικασία βάσει της συνθήκης της ε, Λισαβόνας κατεχώρηση, δεν θα πρέπει να ξαναλέμε επιτροπολογία. Να λέμε πράξη κατεχώρηση λοιπόν. Λοιπόν, πρέπει να ξεσυνηθίσουμε. Τα υγρά λοιπόν παραμένουν ως ήταν, διότι είχαν τύχη επεξεργασία από το κάτω από το παλιό σύστημα, ενώ τώρα έχουμε το νέο σύστημα της Λισαβόνας. Εντάξει. Uh, στα διάφορα. Οι συντονιστέ συζήτησαν μια ιδέα του κύριου Κράμερ για μια συζήτηση για τον τουρισμό, να οργανώσουμε μια τέτοια συζήτηση και συμφωνήσαμε. Για το τρίτο πακέτο σιδηροδρόμων τώρα, όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών και πάλι εδώ ε, ενέκριναν πρόταση που έγινε για να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα έγγραφο όσον αφορά την εφαρμογή του τρίτου πακέτου σιδηροδρόμων και ιδιαίτερα όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρόμων γιατί δεν ακολουθούν πάντα την ίδια γραμμή οι ισοδρομικέ εταιρείε και ζητήσαμε η Επιτροπή να μας ετοιμάσει ένα έγγραφο από αυτού. Όσον αφορά τώρα τις προτεραιότητες για το 2011 στον προπολογισμό, τι δημοσιονομικές, επειδή η προθεσμία είναι πολύ σύντομη από πλευρά τη Επιτροπή Προπολογισμών για τι τροπολογίε 25 Φεβρουαρίου είναι, ο αντιπρόεδρο Ρίκε έχει ετοιμάσει μια σύσταση, με επιστολή σύσταση Προ τον εισηγητή της, των προπολογισμών υπογραμμίζοντα την ανάγκη για του σιδηροδρόμους. Και ο κύριο Ρίκη προτείνει μια συνάντηση ε, με τους σκιώδεις, ώστε μετά να υποβληθούν τροπολογίες. Οπότε παρακαλώ τους σκιώδεις να έρθουν σε επαφή με τον Αντιπρόεδρο. Ξέρω ότι είναι μια κάπως ξεχωριστή διαδικασία, αλλά αυτό είναι γιατί η προθεσμία Τη Επιτροπή Προπολογισμών για τροπολογίε. είναι τόσο σύντομη. Βλέπετε άλλαξε η διαδικασία με τη Λισαβόνα και γι' αυτό αλλάζουν πολλά άλλα επίση. Το επόμενο είναι η συνεργασία μας με τον Επίτροπο Κάλλας. Ναι, ναι, θα ψεφίσουμε, συνάδελφοι, εντάξει. Περιμένετε λίγη υπομονή. Οι συντονιστές λοιπόν ανέκριναν πρόταση δικιά μου για μια πρώτη συνάνταση με τον Επίτροπο Κάλλα στις 9 Μαρτίου στο Στρασβούργο, οι συντονιστές δηλαδή, για να συζητήσουμε λιγάκι τα αποτελέσματα του άτυπου συμβουλίου που θα λάβει η χώρα στη Λαπερούνα και στην Μαδρίτη. Επίσης όμως αποφασίσαμε ότι θα ήταν καλό να έχουμε συναντήσεις τακτικά. Μετά από συνεδριάσεις του Συμβουλίου δηλαδή να έρχεται ο Επίτροπος, στου συντονιστές και να μας λέει τι έγινε. Και μετά οι συντονιστέ εννοείται θα ενημερώνουν όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής για το τι έχει συμβεί. Αυτά όσον αφορά τη συνάντηση των συντονιστών. Εκτό αν οι συντονιστέ ε, θέλουν κάτι να προσθέσουν, μπορεί και κάτι να ξέχασα. Έτσι κι αλλιώ είχαμε τόσα πολλά στην ημερήσια διάταξη που μπορεί να έχω ξεχάσει κάτι. Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι. Έτσι, συμφωνείτε κι εσεί, Ωραία. Αν συμφωνείτε, έχει καλώς και τότε α περάσουμε στις ψηφοφορίε. Εντάξει, σας ευχαριστημένοι τώρα που αρχίζουμε την ψηφοφορία. Μπράβο. Ευχαριστώ που ήσασταν τόσο υπομονετικοί μαζί μου. So. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Πρώτον, δική μου έκθεση για Σχέδιο έκθεση λοιπόν όσον αφορά πρόταση απόφαση για κοινοτικού προσανατολισμού για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Υπάρχουν διάφορε τροπολογίε. Ξεκινάμε με την τροπολογία αριθμό 6 τη κυρία Τικάου. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Ετρολογική σκέψη 19, τροπολογία αριθμό 1 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σκεπτικό τώρα 19α, τροπολογία 3, Κράμερ και Λίχτεμπέργκερ, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 2 έχει αποσυρθεί. Ε, τη λογική σκέψη 20, τροπολογία 4, Σίμψον, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τροπολογία 5 καταπίπτει συνεπώς ε, νομοθετική πράξη. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Οπότε ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εντάξει κύριε Βάκη, έχετε βάλει σωστά την κάρτα σας. 39 ψήφισαν, μέσα με τον κύριο Βάικ. 39 υπέρ, καμία κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Hang όχι, όχι, δεν θέλω να καμαρώσω. Λοιπόν, τώρα το κείμενο νομοθετικού περιεχομένου ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Κάποιος εδώ κάνει σαν Λοιπόν, 37 υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ποτέ δεν είχα τέτοια ομοφωνία σε έκθεσή μου. Τι καλά. Επιτέλους. Just let me bask in the ε, επιτρέψτε μου λιγάκι και εγώ να πενέψω τον εαυτό μου, να καυχηθώ. Επόμενο θέμα. Θα τα πάει εξίσου καλά. Είναι η έκθεση του κυρίου Ελ Καντραουή για σχέδιο γνωμοδότησης για την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Είναι η οδηγία που αφορά την οργάνωση λοιπόν του χρόνου εργασίας των εκτελών των κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Καταρχήν, 1α, τροπολογία αριθμός 6 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Με ελέγξουμε. Εντάξει, θα ελέγξουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Ψήφισαν 39, 18 υπέρ, 20 κατά, μία αποχή. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30, Κρός και Γένσεν. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές θα ελέγξω. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά προτιμώ να το ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 22 κατά. Δύο αποχές. Απορρίπτεται λοιπόν. Άρθρο 1, σημείο 1, αλφα, αλφα νέο. Τροπολογία 31, Γρός και Γένσεν. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7 έχει αποσυρθεί. 32 τώρα του κυρίου Ελκαντραουή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίπτεται και αυτή, αλλά να ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 16 υπέρ, 20 κατά. Δύο αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Γρός Γένσεν. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε. 8. Ψηφίζουμε την 8. Πέρα τη ψηφοφορία. 19 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. Δεν έχουμε αποχές. 9 τώρα του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε πάλι παρακαλώ, συνάδελφοι. Τροπολογία 9 λοιπόν του εισηγητή. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 18 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ίδιο νομίζω είναι το αποτέλεσμα, αλλά ας το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 20 κατά. Βλέπετε, όντως χρειαζόταν να ελέγξουμε. Άρθρο 1, σημείο 2, τροπολογία 11 του εισηγητή. Υπέρ παρακαλώ. κατά αποχές θα το ελέγξουμε αν και νομίζω ότι εγκρίνεται ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 11 ψηφίζουμε πέρα της ψηφοφορίας 19 υπέρ 19 κατά μία αποχή απορρίπτεται δηλαδή Τη κυρία Λίχτεμπερ τώρα, η τροπολογία 34. Ψηφίστε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 35. Γκρό. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 12. Του συγητή. Υπέρ. κατά αποχές θα ελέγξουμε παρακαλώ. Είναι η 12 λοιπόν του συγγετή. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες; 18 υπέρ, 21 κατά, μια αποχή απορρίπτεται. 36 τώρα του κυρίου Ελκαντροή υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 37 του κύριου Ελκαντράουι υπέρ κατά αποχές θα την ελέγξουμε αυτήν παρακαλώ 37 λοιπόν ελέγχουμε ψηφίστε ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι τέλος της πληροφορίας 18 υπέρ, 22 κατά. Αλλιώς θα είχα πρόβλημα. Λοιπόν, 18 υπέρ, 22 κατά. Απορρίπτεται. 38 είναι η επόμενη του κυρίου Ελκαντραουή. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Θα αλλάξουμε και για αυτή την τροπολογία, παρακαλώ. 38 λοιπόν, ψηφίστε. Τέλος της προφορίας. 20 υπέρ, 21 κατά. Απορρίπτεται. Επόμενη τροπολογία της κυρίας Βόρτμαν Κόλλη, 39. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Τροπολογία 39. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα. 39 λοιπόν, ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 20 υπέρ 20 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 τώρα του συγκητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 της κυρίας Λίχτεμπεργκερ. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για τις 40. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 23 κατά. Καμία αποχή. Απορρίπτεται. Τώρα, 13, 15, 16 και 17 έχει ζητηθεί να τις ψηφίσουμε μαζί, αν μπλοκ. Υπέρ παρακαλώ όλων αυτών. Κατά Θα τα ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνονται, αλλά να ελέγξουμε καλύτερα. 13 με 17 υπέρ. Ε, ψηφίστε μάλλον ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 20 υπέρ, 21 κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται όλες αυτές. Άρθρο 1, σημείο 12 τώρα. Πρόκειται για τροπολογία 18 του εισηγητή. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Γκρός και Γένσεν. Εδώ έχει ζητηθεί προφορική τροπολογία. Νομίζω ότι την έχετε. Υπάρχει καμιά αντίρρηση για την προφορική αυτή τροπολογία. Εφόσον όχι, ψηφίζουμε τότε με την τροποποίηση αυτή την προφορική την τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το ελέγξουμε. Πρόκειται για την τροπολογία 19 με την προφορική τροποποίηση. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 23 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται. Να και μια τροπολογία που εγκρίνεται. Σκεπτικό 4α, τροπολογία 20, Βόρτμαν Κόλ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 της κυρίας Τικάου, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμός 1 του εισήγητη έχει αποσυρθεί και έχει αντικατασταθεί από τροπολογία 22 Ελκαντραουή υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το λέξουμε παρακαλώ. 22. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 22 κατά. Μία αποχή. Απορρίπτεται. 23 της κυριαστικά υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. 24. Τροπολογία 24. Εδώ έχει ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς. Έτσι, ξέρετε πώς είναι. Πρώτο τμήμα. Μέχρι το κανονισμός 561 κάθετος 2006 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Πρώτο τμήμα λοιπόν της τροπολογίας 24. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 15 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. να το ελέγξουμε καλύτερα. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα δούμε. Δεύτερο τμήμα λοιπόν, τη 24, ξεκινάει η ψηφοφορία, ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 16 πέρι 23 κατά, μία αποχή απορρίπτεται. Επόμενη τροπολογία είναι 25 της κυρίας Βόρτμαν Κόλ και πάλι έχει ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία από το ECR. Πρώτο τμήμα μέχρι εκεί που μιλάει για την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά τις οδικές μεταφορές. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα. Από εκεί που ξεκινάει ότι είναι για το κοινό συμφέρον. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα καλύτερα. Δεύτερο τμήμα λοιπόν της τροπολογίας 25. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 20 κατά, 2 αποχές. Απορρίπτεται. 26 είναι η επόμενη, γιατί δεν έχει αποσυρθεί και έχει αντικατασταθεί από την 26. Λοιπόν, 26 ελκαντροή υπέρ. κατά αποχές να ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε καλύτερα για την 26. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 21 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 του εισηγητή υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 έχει αποσυρθεί, 27 τώρα που την αντικαθιστά το κύριο Λικαντραή και Λέχτφριντ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 Ελκαντραουή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 Ελκαντραουή υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ αυτή την τελευταία. Τροπολογία 5 λοιπόν του εισηγητή. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 21 κατά, μία αποχή. Απορρίπτεται. Και τώρα ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία, σχέδιο γνωμοδότηση, αλλά προηγουμένω ο κύριο Ελκατραουή θέλει κάτι να πει. Σαΐτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όντω, ε, θα έλεγα ότι είχε περισσότερη αγωνία η ψηφοφορία από ό,τι περίμενα. Πάντω υπάρχουν διάφορα σημεία στην έκθεσή μου που δεν έχουν περάσει. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να στείλουμε την γνωμοδότηση αυτή στην αρμόδια επί της επιτροπής, στην Επιτροπή Απασχόλησης. Οπότε θα έλεγα να μην στηρίξουμε την γνωμοδότηση αυτή κάτω από τις συνθήκες αυτές. Μάλιστα. Ε, συστήνει απόρριψη της ε, έκθεσής του βασικά ο εισηγητής. Εσείς τι έχετε να πείτε. Σύμφωνα απολύτως με τον. Δηλαδή, καταλαβαίνω απολύτως αυτό που θέλει να πει ο συνάδελφος. Όμως πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση οι πολιτικές ομάδες ψήφισαν κατά τη βούλησή τους και επομένως θα πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία. Αργότερα θα προσπαθήσουμε να δούμε εάν τα πράγματα είναι αρκετά όρημα έτσι ώστε να φτάσουμε σε σε ένα συμβιβασμό, πράγμα το οποίο δεν ήταν δυνατόν τώρα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε άλλωστε και την γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, ε, Απασχόλησης, ε, τουλάχιστον έχουμε τις αιτιολογικές σκέψεις. Ναι, ναι. Θα ψηφίσουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Ακούσατε την σύσταση του εισηγητού, ακούσατε και την απάντηση του Μάθιους Γκρός και επομένως επαφίεμαι σε εσά, το αφήνω σε εσά. αρχίζει η τελική ψηφοφορία. Has everybody voted? Εψήφισαν όλοι. Άρα πέρα της ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 20 κατά, μία αποχή. Επομένως απορρίπτεται. Προχωράμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ α, που προείσταμε μια τέτοια αποφασιστικής επιτροπής. Λοιπόν, το επόμενο θέμα, απαλλαγή για την εφαρμογή του Γενικού Προϋπολογισμού για το έτος 2008-2009 για το 2008. Ε, μιλάμε πρώτα για την ΕΠΣΟ. Έχουμε δύο τροπολογίες από την κυρία Γιάλα Σέντερ. Ε, τροπολογία 1 παράγραφος 5 υπέρ. Είμαστε στην ΕΜΣΑ. Η συγκήτρια είναι η κυρία Γένσεν. Το βρήκατε, πολύ ωραία. Παράγραφος, ε, τροπολογία 1, παράγραφος 5, τα είπα ανάποδα. Ο πρόεδρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2, παράγραφος 6, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Α, στο δικό σας κατάλογο είναι άλλη σειρά. Εν πάση περιπτώσει είναι η ΕΜΣΑ πάντως. Τελική ψηφοφορία για την έκθεση Γέννησεν επί της ΕΜΣΑ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 34 υπέρ 3 κατά 2 αποχές. Επομένως εγκρίνεται. Μπράβο κυρία Γέννησεν. Συγχαρητήρια. Ε, δεν ήταν τόσο αποφασιστικό το αποτέλεσμα όσο επί της δικής μου εκθέσεως. Πρέπει να τα λέμε αυτά, λέει ο πρόεδρος, αλλά εν πάση καλά πήγατε κι εσείς. Τώρα, όσον αφορά τον Οργανισμό Ασφάλειας ε, Πολιτικής Αεροπορίας, το βρήκατε. Ναι, άλλαξα λίγο τη σειρά. Παράγραφος 4, τροπολογία 1 της κυρίας Αγιάλα Σέντερ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 επί της παραγράφου 5 της κυρίας Γένσεν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 επί της παραγράφου 6 της κυρίας Γένσεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 της κυρίας Αγιάλα Σέντερ επί της παραγράφου 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επί της παραγράφου 7, τροπολογία 5 του κυρίου Μπαλσάιτης, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για την Ιάσα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. Επόμενο, απαλλαγή για τον ERA, γιατί είναι για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Δύο τροπολογίες έχουμε, του κυρίου Ρικέ. Τροπολογία μη 1, της, επί της παραγραφού 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, επί της παραγράφου 6, πάντα είναι τροπολογία του κυρίου Ρικέ, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται τελική ψηφοφορία για τους σιδηροδρόμους. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 34 υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές, επομένως εγκρίνεται. απαλλαγή για το Σέζαρ της κυρίας Γένσεν. Έχουμε μία τροπολογία του κυρίου Μπαλσάιτης, ε, η οποία απεσήρθη. Όμως, επομένως, τελική ψηφοφορία για το Σέζαρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 34 υπέρ, 2 κατά, 1 αποχή και επομένως εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Γένσεν για την έκθεση αυτή. Έχουμε επίσης ε, την απαλλαγή για τον Γενικό Προϋπολογισμό 2008, τμήμα 3, παράγραφος 5, τροπολογία 1 του κυρίου Κράμερ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Υπάρχει η τροπολογία 2 της κυρίας Σέντερ, ε, ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα από το regrets ε, λυπάται μέχρι of tourism, του τουρισμού. Πρώτο τμήμα λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα καλωσορίζει μέχρι το τέλος υπέρ κατά αποχές. Το δεύτερο τμήμα παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση. Στο δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 2 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 17 κατά, 2 αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 του κυρίου Κράμερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία όσον αφορά την ε, απαλλαγή για το τμήμα 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 34 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή, επομένως εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Γιάλα Σέντερ. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Which is my own report είναι επόμενη η δικιά μου έκθεση. Ακούω εδώ πολύ φασαρία. Okay. I think in, in future colleagues I'm going to get my coffee prior to a long because it's not... Ε, λοιπόν, νομίζω πάντως ότι την επόμενη φορά θα πίνω τον καφέ μου πριν ξεκινήσουν οι ψηφοφορίε, γιατί τώρα πώ να τον πιω που έχει παγώσει. Okay, colleagues, the next item on the agenda is... Το επόμενο σημείο λοιπόν η αφορά τη, τα, ε, τον εξοπλισμό ε, τον μεταφερόμενο μάλλον εξοπλισμό ε, υποπίεση. Νομίζω ότι το πρώτο που μπορώ να πω ξεκινώντας είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο θέμα αφορά τα διάφορα, ε, τους διάφορους τρόπους μεταφοράς, κυρίως αερίων και στόχος ε, αυτής της οδηγίας για τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υποπίεση είναι έτσι ώστε να ε, γίνει ασφαλής η μεταφορά ε, των αερίων αυτών χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά που θα διέρχεται το, το φορτηγό, το βιτίο από κάθε χώρα να χρειάζεται ξεχωριστή άδεια. Ε, πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά τεχνικό, όπως μπορείτε άλλωστε να το φανταστείτε. Και ε, βεβαίως η ουσία της αλλαγής του περιεχομένου δεν τίθεται εδώ. Απλώς θέλουμε να αποσαφηνίσουμε ε, τα στάνταρ τα οποία <clears throat> υπάρχουν στις διάφορες χώρες. Η αναθεώρηση αυτή εκρίθη απαραίτητη λόγω των πολυπληθών αλλαγών της ε, νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια και βεβαίως ε, και σε συνδυασμό με την εναρμόνιση των διεθνών κανονισμών όσον αφορά ακριβώς τη διαθέτηση των λεπτομεριών αφορά τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υποπίεση. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει διεθνή συμφωνία επί του θέματος. Οι τροπολογίες περιλαμβάνουν την αποσαφήνιση του, του ορισμού του μεταφερόμενου εξοπλισμού υποπίεση και αναφέρεται επίσης στον τρόπο πρακτικής εφαρμογής των αρχών. Επίσης περιέχει αποσαφήνιση του γεγονότος ότι δεν χρειάζεται βεβαίωση συμβατότητας ε, ε, σε επίπεδο περιφερειακό ή εθνικό τις ε, τροπολογίες ε, τις οποίες έχω υποβάλει φαίνεται ότι την χάνουν τη συμφωνία του Συμβουλίου γιατί έχω μιλήσει με αυτούς ε, και όσον αφορά την Κομισιόν επίσης θεωρεί ότι ε, ήταν ε, καλές και προς τη σωστή κατεύθυνση οι τροπολογίες μου. Όσον αφορά την επιτροπολογία ή αν θέλετε πράξη κατεχώρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει η επιτροπολογία στο πούμε τώρα, είναι ότι πρόκειται για μια ε, θεσμική, διαθεσμική συμφωνία επί των νέων προνοιών αυτής, αυτού του κανονισμού. Και εντωμεταξύ έχουμε και την μας, το δικό μας σχέδιο έκθεσης, το οποίο περνάει από τις νομικές υπηρεσίες ε, του Κοινοβουλίου ε, και που θα δώσει το δικό μας στίγμα όσον αφορά το θέμα αυτό. Ε, καλό θα ήταν να έχουμε την απόφαση από τις τροπολογίες σε πρώτη ανάγνωση. Βεβαίως ελπίζω ότι δεν θα υποβληθούν περαιτέρω τροπολογίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε με το θέμα αυτό σε πρώτη ανάγνωση. Αυτά όσον αφορά την έκθεσή μου. Ελπίζω ότι πλέον αποσαφήνισα το πεδίο, το αντικείμενο αυτής της έκθεσης προσπαθούμε να έχουμε ένα εναρμονισμένο σύστημα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και που βεβαίως ε, θα ε, ταυτίζεται και, με, και θα ευθυγραμμίζεται και με τις διεθνείς ε, συμφωνίες όσον αφορά τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υποπίεση. Για το ΕΛΚ ο κύριος Κόφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ εξ του ΕΛΚ και να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή σας εργασία. Επίσης θα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή για την πρωτοβουλία σας. Είναι πολύ τεχνική αυτή η έκθεση βέβαια, αλλά εγώ χαιρετίζω τους επιδιωκόμενους στόχους. Μεγαλύτερη λοιπόν ασφάλεια είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιτευχθεί και στα κράτη-μέλη και μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις μεταφορές. Αυτό δεν σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε το νομικό πλαίσιο, απλώς να ξεπεράσουμε τις αντιφάσεις που υπάρχουν μεταξύ υφισταμένων οδηγιών και διεθνών ρυθμίσεων για τα θέματα αυτά και να υπάρξει και μία καλύτερη προσαρμογή με την, ε, προς την οδηγία που είχαμε εγκρίνει πριν από δύο χρόνια για τη μεταφορά επικινδύνων ε, αντικειμένων και υλικών στο δρόμο, στους σιδηροδρόμους και στις εσωτερικές υδάτινες οδούς. Υπάρχει λοιπόν και η ανάγκη να υπάρξει μια πιο αυστηρή αντιμετώπιση των παραβάσεων όπως επιτυγχάνεται με την τρέχουσα οδηγία. Έρχομαι τώρα στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και εδώ αναφέρεται στους, ε, στα δοχεία τα οποία μπορούν να αναγεμίζονται. Δεν έχω καταλάβει γιατί γίνεται αυτή η διάκριση σε σχέση με τα κοντένες, με τα δοχεία αυτά. Ο κύριος Στέρξ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, βεβαίως εξ ονόματος κυρίου Μάισνερ, ο οποίος ασχολείται με το θέμα αυτό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε για αυτό το τόσο τεχνικό θέμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια ρύθμιση για την Ευρώπη, η οποία να συνάδει με τους διεθνείς κανόνες. Το θέμα της ε, ασφάλειας είναι βέβαια κάτι που ποτέ δεν μπορούμε αρκετά να τονίσουμε. Και πέρυσι στο Βιαρέτζο θα θυμόσαστε στην Ιταλία που άνοιξε ένα τέτοιο τάνκερ και κάπου δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν. Νομίζω λοιπόν ότι οι προδιαγραφές πρέπει να είναι πολύ ψηλέ. Συμφωνούμε απόλυτα λοιπόν με την γραμμή που ακολουθείτε εσείς Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Η Κομισιόν θα ήθελε να λάβει το λόγο για το θέμα Ο κύριος Πασπαρέλη. Κύριε Πασκαρέλη, αν μπορείτε να αντιμετωπίσετε και το πρόβλημα που έθεσε ο κύριος Κοκ, γιατί εγώ δεν έχω γνώση του θέματος. Αυτό είναι μια νέα εξέλιξη. Πράγματι, λέει ο κύριος Πασκαρέλη να απαντήσω πρώτα στον κύριο Κόκ και θέλω να το διαβεβαίωσω ότι οι μη αναγωμούμενοι εξοπλισμοί υποπίεση καλύπτονται απόλυτα από αυτή την οδηγία, αλλά, αλλά επειδή δεν μπορεί να υπάρξει εκ νέου ε, γέμισμα αυτών των δοχείων, δεν, δεν έχει νόημα το αν έχουν τμήματα τα οποία μπορούν να αποσυνδεθούν ή όχι. Από τη στιγμή που χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά, μετά απορρίπτονται. Οπότε δεν χρειάζεται να περάσουν πάλι τη διαδικασία έγκριση. Επομένω, η ανησυχία σα έχει ληφθεί υπόψη. Εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα εξαρτημάτων τα οποία μπορούν να περασουμε παλι τη διαδικασια εγκριση επομενω η ανησυχια σα εχει ληφθει υποψη εφοσον δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί όταν έχουμε ένα εξοπλισμό ο οποίο χρησιμοποιείται μονάχα άπαξ, τότε μετά το άπαξ τον πετάμε. Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνολικότερα, εγώ δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που είπε ήδη ο εισηγητή, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους ομιλητές που έλαβαν το λόγο. Νομίζω ότι έχουν <clears throat> περιγράψει την κατάσταση επακριβώς. Το μόνο το οποίο εγώ θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι η έγκριση αυτού του κειμένου από τις ε, νομοθετικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδοκάται αδειμόνως από την βιομηχανία, από τους επαγγελματικού κύκλους γιατί είναι μια, θα είναι μια απάντηση στις τροποποίησεις που έχουν επέλθει στο, στο νομικό πλαίσιο. Η Κομισιόν μπορεί να δεχτεί όλες τις τροπολογίες του εισηγητού με την προϋπόθεση ότι προς το παρόν θα συμφωνήσουμε να διαφωνούμε σε σχέση με τις κατεχώρησης πράξεις αναμένοντας πάντα να υπάρξει μια συνολική επίλυση αυτού του προβλήματος σε διαθεσμικό επίπεδο. Υπάρχει και κάποιο κατεπήγον για να υπάρξει αυτή η συμφωνία για το κείμενο αυτό από τις νομοθετικές αρχές, διότι τα κρατημέλη έχουν επομιστεί ορισμένες διεθνείς υποχρεώσεις στο ευρύτερο πλαίσιο της μεταφοράς επικινδύνων αγαθών, <clears throat> ιδιαίτερα για δοχεία υποπίεσης, Όλα αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου του 2011 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Επομένω, τα κράτη-μέλη χρειάζονται κάποιο χρόνο για να μπορέσουν να μεταγράψουν και να εφαρμόσουν την οδηγία. Όσο πιο γρήγορα, τόσο πιο καλύτερα. Όσο πιο γρήγορα έχουμε λοιπόν μια συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, τόσο πιο εύκολο θα είναι για τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτό το νέο νομοθέτημα. Ευχαριστώ πολύ και ο Μπράιν προβλέπεται η προθεσμία για τις τροπολογίες 25 Μαρτίου, σύγχρον Φεβρουαρίου. Οι τροπολογίες θα εξεταστούν στις 22 Μαρτίου, θα ψηφίσουμε στις 23 Μαρτίου και αν θέλει ο Θεός στην Ολομέλεια μέσα στον 2010, τον Απρίλιο 2010. Ε, πρόκειται για πρώτη ανάγνωση φυσικά, αλλά σας δίνω ποιο είναι το, το χρονοδιάγραμμα για το θέμα αυτό. Εντάξει, εάν είσαστε όλοι ευτυχείς, μπορούμε να περάσουμε στο σχέδιο έκθεσης για το μέλλον των μεταφορών. Κύριος Μάτιου Γκρός έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα θα λάβει χώρα μια πρώτη συζήτηση για αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδησιητές αλλά και όλους τους συναδέρφους οι οποίοι έχουν προσφέρει σημαντικές προτάσεις και ιδέες και μου έχουν αναφέρει σημεία ενδιαφέροντό τους. Εμεί προσπαθήσαμε λοιπόν να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το έγγραφο αυτό. Δεύτερον, εκ προημίου θέλω να σας πω ότι αυτό παραμένει σε επίπεδο, το έγγραφο αυτό παραμένει σε επίπεδο εγγράφου εργασία και ίσως θα πρέπει να το δούμε σαν μια μορφή προκατακτικής αντιμετώπισης για τη Λευκή Βίβλο. Επομένως δεν χρειάζεται να μπούμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, πρέπει να παραμείνουμε μονάχα στο επίπεδο μερικών βασικών ιδεών. Οι αιτιολογικές σκέψεις και το σύνολο του εκτελεστικού του κειμένου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν σύνολο. Αν κάτι δεν περιλαμβάνεται σε ένα τμήμα του εγγράφου θα το βρείτε στο άλλο τμήμα του εγγράφου και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή διάρθρωση του κειμένου. Εγώ θα ήθελα τώρα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένα σημεία. Προφανώς ενδιαφερόμαστε ως Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού να αντιμετωπίσουμε τα θέματα μεταφοράς ως ουσιώδη στοιχεία της ανάπτυξης των περιφερειών, των κρατών μελών και τη Ευρώπη, και να υποστηρίξουμε ιδιαίτερα και να υπογραμμίσουμε το ρόλο των μεταφορών διότι οι δυνατότητες μεταφορών εξασφαλίζουν και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα των κρατών και των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ο τομέα των μεταφορών και σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο απασχόληση παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. Το τρίτο σημείο αναφέρει ότι προφανώς οι μεταφορές έχουν και μεγάλη επίπτωση στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των πολιτών και αυτό το έχουμε ήδη αναφέρει και καταγράψει σε προηγούμενα προγράμματα και εκθέσεις. Το πακέτο για την κλιματική αλλαγή παραμένει για μας ένα σημαντικό σύνολο στοχοθεσιών μέσα στα πλαίσια του ορόσημου του 20, 2020 και εμείς θεωρούμε ότι για τα θέματα των μεταφορών σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να παραμείνουμε η επί της ουσίας επιτροπή. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν άλλες επιτροπές, αλλά πιστεύουμε ότι ό,τι έχει να κάνει με τις μεταφορές θα πρέπει να παραμείνει στα πλαίσια της δικής μας επιτροπής. Η συνεκτικότητα στην αντιμετώπιση για μένα είναι κάτι απαραίτητο σε ό,τι αφορά την γενική προβληματική των μεταφορών. Οι μεταφορέ δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ω ένα μεμονωμένο πεδίο του εμπιστητού. Έχουν μια άμεση επίπτωση στο περιβάλλον οι μεταφορέ, αλλά επίση και στα θέματα τα κοινωνικά, τη απασχόληση, την σύνολη οικονομική πολιτική σε διάφορε χώρε. Και γι' αυτό το λόγο εμεί έχουμε επιμείνει να υπάρξει η σωστή περιχαράκωση των αρμοδιοτήτων μας ως Επιτροπής ώστε να μην καταληφθούν όλα αυτά τα στοιχεία από άλλες πτυχές όπως είναι παραγωγής η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να παραμείνουν εστιασμένα στην Επιτροπή Μεταφορών για την επίτευξη σημαντικών στόχων. Για μένα είναι σημαντικό να υπάρξει μια σωστή καταγραφή των στόχων μας. Η οικονομική ανάπτυξη και η ανάπτυξη των ε, περιφερειών τα επόμενα 10 ή 20 χρόνια θα πρέπει να εξυπηρετηθούν με σαφέστερη στοχοθεσία στον τομέα των μεταφορών και αυτό προσπαθώ να επιτύχω και στο έγγραφο αυτό. Υπάρχουν τώρα συγκεκριμένες προτάσεις. Ε, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ε, κινητικότητα στις πόλεις γιατί 80% του πληθυσμού αύριο θα ζει στις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητο επίσης να δώσουμε έμφαση στην πολυτροπική ε, στις πολυτροπικές μεταφορές, ιδίως στις πόλεις, με ενίσχυση των δημοσίων μέσων μεταφοράς. Αυτό θα είναι λοιπόν ένα εγχείρημα το οποίο θα εξασφαλίσει και το μέλλον των πόλεων. Επίσης είναι γνωστό ότι αυξάνεται η ζήτηση στον τομέα των μεταφορών και αυτό οδηγεί και σε μία ε, μορφή ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Αλλά δεν πρέπει να το δούμε μονάχα σε θέμα ανταγωνιστικότητος μεταξύ των τρόπων μεταφοράς, θα πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ των τρόπων μεταφοράς για να ευνοήσουμε την ε, αποτελεσματικότητα. Η διατροπική λοιπόν ε, οι διατροπικές μεταφορές έχουν μια μεγαλύτερη αποδοτικότητα όχι μονάχα σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Διοξίδιο του άνθρακος, η απανθρακοποίηση είναι αυτός ο νεολογισμός, είναι ένας σημαντικός λοιπόν στόχος τον οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τον επιτύχουμε σε διάφορα επίπεδα σε ό,τι αφορά το μείγμα ενέργειας που χρησιμοποιούμε αλλά νομίζω εδώ και τα μέτρα τιμολόγησης ανήκουν στις προσπάθειες οι οποίες θα ευνοήσουν τη μείωση της χρήσης άνθρακος η εσωτερικοποίηση του κόστους του, της χρήσης του άνθρακα θα πρέπει να είναι και αυτό ένα τμήμα του θέματος το οποίο αντιμετωπίζουμε και φυσικά θα πρέπει να έχουμε και εκεί κίνητρα οικονομικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο πρόσφορα τα οικονομικά κίνητρα από ότι τα οι κυρώσεις, διότι οι κυρώσεις ουσιαστικά δεν οδηγούν σε μια τροποποίηση της συμπεριφοράς και δεν μας οδηγούν να αποφύγουμε αυτά που θέλουμε να αποφύγουμε. Η αποτελεσματικότητα λοιπόν στις διατροπικές ε, μεταφορές είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Να χρησιμοποιούμε λοιπόν τον καλύτερο τρόπο μεταφοράς, ο οποίος σε κάθε περιοχή είναι ο πιο πρόσφορος επί τη βάση των κριτηριών που αναφέρθηκαν προηγουμένω. Επίση, η συμπλήρωση τη εσωτερική αγορά θα πρέπει να παραμείνει στο στόχαστρό μας και αυτό περιλαμβάνει διάφορες πτυχές. Πρώτα απ' όλα αυτά τα οποία αποφασίζονται θα πρέπει να εφαρμόζονται και στην πράξη. Θα πρέπει στο μέλλον να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο να υπάρχει αποτελεσματικότητα στην νομοθεσία την οποία εμείς εγκρίνουμε και μετά στο να εφαρμόζεται αποτελεσματικά και να υπάρχει εποπτεία και παρακολούθηση να δούμε αν υπάρχουν καθυστερήσεις, στρεβλώσεις οι οποίες μπορούν να προκύψουν από λανθασμένη εφαρμογή και επίσης στον τομέα των ε, μεταφορών, παραδείγματος χάρη στο συνδεδομικό τομέα, να δούμε αν πράγματι η φιλελευθερωποίηση αυτού του τομέα επιτυγχάνει τους ε, στόχους για τους οποίους έχει δημιουργηθεί. Η κατάρτιση εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία, γιατί απαιτείται να υπάρχει κατάλληλη ε, πιστοποίηση και δημιουργία προσόντων των εργαζομένων στους τομείς μεταφοράς εγώ νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε και κέντρα αριστείας στα διάφορα κράτη-μέρη. Δεν αρκεί μονάχα να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, αλλά δεν δίνουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να διαπιστώσουν ότι πράγματι η κατάρτιση σε ορισμένες χώρες είναι αποτελεσματική προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ των διαφορετικών κέντρων κατάρτισης. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε παραγωγή χάρη μια αντιμετώπιση που λέει ότι σε δύο ή τρεις εβδομάδες δίνονται τα διπλώματα οδήγηση ενώ αλλού χρειάζονται τρεις μήνες. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν και κάποια, ε, κάποια ενοποίηση στις διαδικασίες αυτές. Για τα προγράμματα έρευνα, νομίζω ότι είχαμε μέχρι στιγμή μια καλή εμπειρία και έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικέ προκλήσει σε προγράμματα τα οποία είναι εν εξελίξη. Παραδείγματο χάρη το πρόγραμμα Open Sky, όπου αφορά την ε, <clears throat> ασφάλεια στι εναέρειε μεταφορέ, που είναι και ακρογωνιαίο λήθο σε ό,τι αφορά τις ε, μορφές μεταφορών, όχι μόνο στις εναέριες αλλά κυρίως και στο, στις οδικές μεταφορές. Επίσης οι αποκεντρωμένοι φορείς, είχαμε πολλές συζητήσεις για το ρόλο των αποκεντρωμένων φορέων. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τέτοιους φορείς οι οποίοι θα προσθέτουν αξία σε επίπεδο αποτελεσματικότητας και όχι μονάχα χώρους συζήτησης. Αν λοιπόν οι αποκεντρωμένοι φορείς μπορούν να συμβάλλουν στην ε, ε, ολοκλήρωση και στην ενοποίηση των προτύπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε μπορούν να προσθέτουν αξία οι αποκεντρωμένοι φορείς, ιδίως σε τεχνικό επίπεδο και φυσικά μπορούμε να θέσουμε ερωτήματα όπως το γιατί δεν υπάρχει κανένας φορέας ειδικά για τις οδικές μεταφορές των 75% των μεταφορών γίνονται με οδικό τρόπο. Μπορούν λοιπόν οι αποκεντρωμένοι φορείς να προωθήσουν την έρευνα, να προωθήσουν, να προαγάγουν την ε, ασφάλεια στο δρόμο και να αντιμετωπίσουν ακόμα και τις στρεβλώσεις και τις δυσκολίες οι οποίες παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά την ε, μεταγραφή και την εφαρμογή των οδηγιών σε διάφορα Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για να έχουμε ένα περαιτέρω φορέα μόνο και μόνο για να έχουμε ένα φορέα, αλλά για να καλύψουμε κάποια κενά τα οποία υπάρχουν στον τομέα της έρευνας και της παρακολούθησης της ε, εφαρμογής. Έχω θίξει λοιπόν ήδη τα θέματα της έρευνας και της τεχνολογίας. Νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε πολλά σε ό,τι αφορά την βελτίωση της ε, αποδοτικότητας της ενέργειας, σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια στους δρόμους κτλ. Και επίσης να έχουμε μια καλύτερη αλυσίδα επιμελητίας κατά κάποιο τρόπο σε ό,τι αφορά την μεταφορά των αγαθών. Αυτό είναι, αυτά είναι ζητήματα τα οποία άπτονται της έρευνας. Και τώρα έρχομαι στο λεγόμενο Ταμείο Μεταφορών, μια δική μου πρόταση. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ένα τέτοιο ταμείο μεταφορών. Γιατί όλα αυτά, γιατί αν θέλουμε στο μέλλον να προχωρήσουμε σε μια σοβαρή συζήτηση με τα, με τα κράτη-μέλη για βελτιώσει στον τομέα των μεταφορών, θα δούμε ότι δεν αρκεί μια θεωρητική συζήτηση, πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένα χρηματικά ποσά, γιατί έχουμε αλλαγές από ένα επίτροπο σε ένα άλλο επίτροπο, από μία περιφέρεια σε μία άλλη περιφέρεια αλλάζουν τα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν μία δυσκολία να εφαρμόσουμε χωρίς κάποια συνέχεια τις ε, προτεραιότητές μας. Ένα ταμείο μεταφορών με τα μέσα τα οποία θα θέσει στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορεί να υποστηρίξει πολύ καλύτερα την περιφερειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προχωρήσει προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής. Νομίζω ότι στα πλαίσια των συζητήσεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα για τη νέα μορφή του προπολογισμού θα ήταν μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Και μια δεύτερη πτυχή ενός τέτοιου ταμείου για τις μεταφορές που εγώ θα ήθελα εδώ να υποστηρίξω συνδέεται άμεσα με το, με το θέμα που συζητήσαμε για την Ευρωβινιέτα, για τη λεγόμενο προς προσδιορισμό των εσόδων που θα προέρθουν από αυτή τη βινιέτα. Δηλαδή μπορούμε να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη τα ποσά τα οποία προερχόνται από αυτή τη βινιέτα να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους στόχους, όπως παραδείγματος χάρη προώθηση της κινητικότητας. Αν έχουμε όμως ένα συγκεκριμένο ταμείο όπου τα χρήματα αυτά, όλες, όλες οι πρόσοδοι από τις βινιέτες μπορούν να μπαίνουν σε αυτό το ταμείο το οποίο θα την χάνει συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα είναι υποχρεωτικό ο προσδιορισμό των κονδυλίων αυτών για να αντιμετωπίσουν τι ανάγκε μεταφορών, αυτό θα είναι ιδιαίτερα πρόσφορο. Γι' αυτό το Ταμείο αυτό μεταφορών μπορεί να καλύψει ιδιαίτερα όλε τι ε, μεταφορέ, αλλά συγκεκριμένα θέματα όπω είναι η ένα η εσωτερική υδάτινη δρόμη, οι εναέρες μεταφορές κτλ. Επομένως, ένα τέτοιο στοιχείο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διευρωπαϊκών δικτύων και θα αποτελέσει και ένα χώρο που θα μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Είναι μια παροχή κριτηρίων, μια παροχή κινήτρων μάλλον, για μεγαλύτερη ε, συνεκτικότητα της δράσης μας στον τομέα των μεταφορών. Προσπάθησα λοιπόν μέσα στο εγγραφό να θέσω ορισμένους εφικτούς στόχους και στο παρελθόν έχουμε διαπιστώσει ότι στο παρελθόν, ιδίως στον τομέα των οδικών μεταφορών, όταν, θέτου, όταν θέσαμε μετρήσιμους στόχους και στόχους που μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ε, επίτευξή τους, αυτό ήταν θετικό. Νομίζω λοιπόν ότι οι στόχοι που θα θεσπίσουμε θα πρέπει καταρχήν να είναι στόχοι οι οποίοι θα κάνουν σαφέστε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορατή για τον πολίτη. Δεύτερον, θα θέσουν τα βασικά κατευθυντήρια στοιχεία. Αλλά και τρίτον, θα πρέπει να είναι ποσοτικοποιήσιμοι αυτοί οι στόχοι και θα μετρήσιμοι ώστε να δούμε κατά πόσο προχωρούμε προς τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει στον εαυτό μας. Επομένως, οι στόχοι αυτοί για μένα αφορούν καταρχήν την ασφάλεια στους δρόμους, στις οδικές μεταφορές και μπορούμε εδώ να έχουμε τα στοιχεία τα οποία θα δείξουν κατά πόσο έχουμε βελτιώσει την ασφάλεια. Ο δεύτερος στόχος αφορά την κινητικότητα στις πόλεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι δεν θα έχουμε στόχο για τα 80% των πολιτών που θα ζουν στις πόλεις. Τρίτον, για την αποδοτικότητα της ενέργειας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την ε, επανεξισορρόπηση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Έχετε λοιπόν ένα κατάλογο τον οποίο μπορούμε, μπορείτε να τον επεκτείνετε ή να τον μικρύνετε, να τον τροποποιήσετε, αλλά γενικά εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια σαφή στοχοθεσία γιατί αυτό ευνοεί ιδιαίτερα την εργασία μας και της δίνει μια συγκεκριμένη βάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας λοιπόν και ελπίζω ότι και σε επόμενες εβδομάδες επί τη βάση αυτού του εγγράφου εργασίας θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρός για αυτή την ε, εξαντλητική παρουσίαση. Ο κύριος Αλκαντράου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Η συνάδελφος Μαγδαλένα που είναι σκιώδης εισηγήτρια μου ζήτησε να πω και εγώ μερικά πράγματα. Η έκθεση αυτή φυσικά και είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι η βάση για τη δουλειά μας τα επόμενα χρόνια. Προετοιμαζόμαστε. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προσπάθεια αυτή. Είναι μια καλή βάση για να δουλέψουμε πάνω σε αυτή. Θέτει τα σωστά ερωτήματα, ακολουθεί τη σωστή προσέγγιση που βρίσκω και εγώ ότι είναι αναγκαία. Με πάρα πολλά πράγματα συμφωνώ αλλά ίσως θα επικεντρωθώ περισσότερο σε θέματα τα οποία θα ήθελα να συμπληρώσουμε. Το κόστος για τις μεταφορές. Συμφωνώ με αυτά που λέτε μαζί σας. Εσείς μιλάτε για τις συνδυασμένε μεταφορές, ναι. Εφόσον πρόκειται για μια επιλογή να υπάρχει αυτή η δυνατότητα συνδυασμού των μεταφορών. Να μπορούμε δηλαδή να μεταφερόμαστε σε άλλα μέσα μεταφορά. Να δούμε πώ θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα προ αυτή την κατεύθυνση. Επίση, προτιμάτε και οικονομικά κίνητρα αντί για κυρώσει. Εντάξει. Αν μιλάμε για το εξωτερικό κόστος που θέλουμε να γίνει εσωτερικό, αυτό δεν σημαίνει, ότι θα πληρώνουμε περισσότερα από όσα πληρώνουμε σήμερα, γιατί θα προκύψει επιπλέον κόστος Μερικές φορές οι κυρώσεις είναι αναγκαίες. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα μοντέλο για το κόστος όλων των ε, μέσων μεταφοράς. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να ξεκινήσει. Για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Τώρα για την εσωτερική αγορά. Μιλάτε για άνοιγμα της αγοράς. Εδώ επίσης σίγουρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Για μένα δεν πρέπει να είναι αυτός σκοπό το άνοιγμα της αγοράς, μπορεί όμως να αποτελέσει μέσο επίτευξης στόχων. Λείπει κάτι όμως για την κοινωνική διάσταση και τι ρόλο μπορεί να παίξει η Επιτροπή σε αυτό για να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση. Επίσης όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς ε, οργανισμούς. Το θέμα του τεχνικού συνδυασμού. Εδώ πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια του οργανισμού για τους σιδηροδρόμους. Είδαμε τι έγινε στο Βέλιο. Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι πρέπει να προχωρήσει περισσότερο να ενισχυθεί, να οριμάσει. Ίσως πρέπει λοιπόν να πούμε κάτι και εδώ για ένα πρόγραμμα δράσης υπέρ της κινητικότητας. Πώς μπορούμε να ελέγξουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα αυτά τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά το ΙΤΕΣ, ίσως πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα, να πιέσουμε. Και τέλος, Μεσοπρόθεσμοι στόχοι, ναι, σωστά. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρώπη γενικότερα είναι καλό να θέτουμε στόχους που να μπορούμε να τους πετύχουμε. Εγώ δεν θα μιλούσα για το παράδειγμα που φαίνεται εσείς εδώ. Πρέπει να το δούμε. Αλλά γενικά η προσέγγιση σας είναι σωστή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ μιλάω εκ μέρους της κυρίας Στισμπερκ η οποία είναι σε προεκλογική εκστρατεία στην εκλογική της περιφέρεια. Αυτή είναι εκπρόσωπο εδώ. Καταλαβαίνετε ότι οι προτεραιότητες μερικές φορές δεν είναι να είναι κανείς εδώ. Υπάρχουν και πράγματα σημαντικά στις χώρες μας μερικές φορές. Λοιπόν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για τον τρόπο με τον οποίο έχει συνεργαστεί με τους σκιώδες εισηγητές για να φτάσει σε αυτό το έγγραφο. Θέλω λοιπόν ε, να το τονίσω αυτό. Από εδώ και πέρα, ίσως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι χρειαζόμαστε μια αρκετά ευρία πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στις συζητήσεις που θα έχουμε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για να είναι ισχυρή η θέση μας. Δεύτερον, πρέπει επίσης πολύ συγκεκριμένα θέσεις να υποστηρίζουμε. Και γι' αυτό είναι καλό το κεφάλαιο με τους μετρήσιμους στόχους. Πρέπει να συζητάμε για ποσοστά, για νούμερα, αλλά έτσι κι πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος με ορισμένα πράγματα που να λέμε ότι θέλουμε να τα δούμε με ποσοτική έκφραση. Ξέρω εγώ πόσο, τις 100 μείωση θυμάτων λέω για παράδειγμα. Είναι σημαντικό το κοινοβούλιο να λέει να, αυτή είναι η γραμμή που εμείς θέλουμε να κρατήσουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο εισηγητής πολύ σωστά μιλάει για τις αποτελεσματικές συνδυασμένε μεταφορές. Πρέπει να είναι αποτελεσματική διαφορή τρόπη μεταφοράς. Αυτή είναι η λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την κινητικότητα κάθε μέσο μεταφοράς έχει τα υπέρ και τα κατά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οπότε πρέπει να συνδυάσουμε διαφορετικά μέσα μεταφοράς ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα πλεονεκτήματα. Και το κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να πιέσουμε και να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μεγαλύτερο ρόλο να παίξει. Δεν ξέρω τα κράτη-μέλη πάντα στη θεωρία λένε «Α, ναι, ναι, η Ευρώπη να πληρώσει, ναι», αλλά όταν οι Υπουργοί Οικονομικών ή Δημοσιονομικών ετοιμάζουν τον προπολογισμό, τότε γι' αυτό λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει, να διορθωθεί. Το κεφάλαιο τώρα για τους οργανισμούς είναι σημαντικό. Και χαίρομαι πολύ που μιλάτε και για τον οργανισμό για τις οδικές μεταφορές, γιατί δεν πρόκειται μόνο για τους άλλους τομείς, πρόκειται και για αυτόν. Βρίσκω την επιχειρηματολογία σας πολύ σωστή. Μία ερώτηση έχω να κάνω. Στον κατάλογο με τους στόχους για το διοξίδιο του άνθρακα γίνεται μια σύγκριση με το 2010, ενώ στο πακέτο για το κλίμα ως βάση παίρνουμε ως ε, έτος αναφοράς το 2005. Δεν θα ήταν προτιμότερο να βάλουμε και εδώ το 2005. Μια ερώτηση είναι αυτή. Και δεύτερον ως ομάδα ρωτάμε δεν θα έπρεπε να φροντίσουμε και για αναλλακτικά καύσιμα όσον αφορά τις οδικές μεταφορές, να μιλάμε για το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο. Στο σημείο για τις καινοτομίες ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα προσωπικά θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημασία που δίνετε στην εσωτερική αγορά. Πιστεύω ότι αυτό που λέει και ο Σαΐντ για τη σημασία που έχει η εσωτερική αγορά είναι σωστά. Αλλά τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν εύκολα να μεταφέρουν αρμοδιότητες τους για τις μεταφορές σε ένα άλλο επίπεδο. Ενώ αυτό θα μπορούσε να γίνει και θα έπρεπε. Είτε για το short ship ε, shipping. Εδώ η εσωτερική αγορά έχει να παίξει σημαντικό ρόλο. Αλλά είναι δύσκολο. Είτε όταν μιλάμε για τη χρήση των γλωσσών, για παράδειγμα, βλέπουμε τι πρόβλημα υπάρχει η εσωτερική αγορά όμως μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο σε επίπεδο ρύθμισης αλλά και στη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων ώστε να γίνει πιο εύκολη η καθημερινή διακίνηση εμπορευμάτων. Θα έχουμε πολλές καρποφόρες, πιστεύω, συζητήσεις μεταξύ μας. Η ομάδα μας υποστηρίζει σε γενικέ γραμμές την πρότασή σας και από εκεί και πέρα χρειάζεται παρετέρω συζήτηση για να διευκρινιστούν κάποια επιμέρους θέματα πάνω στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε για ποσοστά, για συγκεκριμένους στόχους, αλλά έτσι κι αλλιώς με αυτή την έκθεση σίγουρα θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λίχτεμπεργκ, εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκρός για την πλήρη και εμπεριστατωμένη έκθεσή του και έχει πολλά θετικά στοιχεία. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια συζήτηση η οποία είναι απαράγραπτη σε σχέση με το μέλλον. Είναι θετική οι στόχοι οι οποίοι τίθενται ε, διότι έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια και συγκεκριμένο τρόπο και πιστεύω ότι είναι και ρεαλιστική αυτή η στόχη του οποίου θέτει ο εισηγητής. Εγώ θα ήθελα όμως μεγαλύτερη σαφήνεια. Συγγνώμη. Με τις υγείες σας κυρία Λιχτεμπερκ λέει ο πρόεδρος για την ε, κίνηση στις πόλεις. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και μια διαφοροποίηση μεταξύ της κινητικότητος ως αναγκαιότητος και ως αξίας. Γιατί η κινητικότητα σημαίνει και μεγαλύτερες μεταφορές και σε πολλές περιπτώσεις ο πολίτης κατανοεί την κινητικότητα μόνο με το αυτοκίνητο στις πόλεις. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διατυπώσεις που θέλουμε να έχουμε. Δεύτερον, επειδή αναφερόμαστε στο μέλλον, δεν θα πρέπει να έχουμε την έννοια της ε, διαφοροποίησης μεταξύ των τρόπων μεταφοράς. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μεν χωριστά τους τρόπους μεταφοράς, αλλά να τονίσουμε ότι αν δεν υπάρξει μια μετατόπιση από τους δρόμους στο σιδηρόδρομο για τη μεταφορά αγαθών αλλά και μέσα στις πόλεις ακόμα δεν θα μπορέσει να υπάρξει η επίτευξη των στόχων. Γιατί αν πρόκειται εμεί να κόψουμε όλα τα δάση στην Βραζιλία για να έχουμε βιοκαύσιμα, τότε δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή η πολιτική. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε με σαφήνεια ότι είναι απαραίτητη μια μετατόπιση των μεταφορών από τις οδικές μεταφορές και αυτό είναι σημαντικό να γίνει στο μέλλον και να αποφευχθεί επίσης και η περιττή μετακίνηση. Αυτό λοιπόν είναι τα θέματα τα οποία έρχονται στο μυαλό μου όταν προσπαθούμε να σκεφτούμε με το μέλλον των μεταφορών. Διότι η μεταφορά μεταφορές έχουν να κάνουν και με τη χωροταξία και με την ολοένα συνεχιζόμενη μετακίνηση των εργαζομένων στις παρυφές των πόλεων. Όλα αυτά λοιπόν έχουν και μία σημασία για μας. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε τέτοιες εξελίξεις οι οποίες συνδέονται με μία ανάπτυξη των μεταφορών. Επίσης, το σημείο 4 βρίσκεται σχεδόν σε αντίφαση με τα θετικά στοιχεία τα οποία τόνισε ο εισηγητής. Εμείς θα πρέπει να κατονομάσουμε με σαφήνεια ότι πρέπει να υπάρξει μια ανακατεύθυνση στον τομέα των μεταφορών και εάν εμείς θέλουμε να επιτύχουμε τους ε, στόχους της κλιματικής αλλαγής και είναι πολύ σωστό που τους υπογραμμίζει ο εισηγητής, αυτό θα απαιτήσει και, σε αλλαγέ, αλλαγές στον τρόπο διαβίωσης και μεταφορών μας. Κάτι ακόμα είχα να αναφέρω για τις θετικές επιπτώσεις των μεταφορών. Στη, στον τομέα των οικονομικών, όμως, στον τομέα της οικονομικής δραστηριότητας θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι μεταφορές στο δρόμο αλλά και εν μέρη και στους σιδηροδρόμους μπορούν να έχουν και αρνητικές επιπτώσεις. Ότι οδηγούν και σε απώλεια ποιότητος ζωής, ότι οδηγούν σε υποβάθμιση της ανθρώπινης υγείας σε πολλές περιπτώσεις και σε ό,τι αφορά τη χωροταξία και την ε, ανάπτυξη των, ε, του, της υπαίθρου οδηγούν ουσιαστικά σε μια απογύμνωση των ε, περιφερειών διότι επιτρέπουν μια υπερσυγκέντρωση της δραστηριότητας της πόλης. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα πρέπει και αυτά να αντιμετωπιστούν σε περαιτέρω συζητήσεις εάν θέλουμε να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση των μελλοντικών προοπτικών. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να επανέλθω στο λεγόμενο modal split, δηλαδή στο χωρισμό των διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Εάν θέλουμε να δούμε πώς θα είναι το μέλλον, θα πρέπει να αποφύγουμε και να αντιμετωπίσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των τρόπων μεταφοράς. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε την φορολογία ορισμένων καυσίμων και να φορολογηθεί και η κυροζήνη. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να προχωρήσουν υπό μορφή φορολογικών μέτρων. Και αυτό είναι μια αίτηση την οποία θέλω να διατυπώσω σαφώς από τη δική μου πλευρά και σας λέω θα καταθέσω και τροπολογίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Βαντάλεν. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε για την ε, έκθεσή σας και για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίσατε κάποιες ε, ιδέες. Μας βρίσκουν σύμφωνους ε, οι ιδέες σας και επομένως συμφωνούμε με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τα πράγματα. Όσον αφορά τώρα τους μετρήσιμους στόχους, χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχετε τα στοιχεία αυτά μέσα, θα πρέπει, αλλά βλέπουμε ότι ε, πρόκειται για εξαιρετικά καλή ιδέα αυτή η μετρήσιμη ε, ε στόχη, αλλά ε, βεβαίως ε, θα πρέπει να δούμε και σε σχέση με την ετήσια εκπομπή ρήπων πώς μπορούμε να έχουμε και εκεί μετρήσιμους στόχους και ποια θα είναι η βάση μέτρησης βέβαια που θα έχουμε. Υπάρχουν ε, και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία με δυσκολεύουν λίγο και θα συμφωνήσω με την ε, κυρία Λίχτεμπεργκερ. Δηλαδή αυτή η διατροπικότητα δεν είμαι βέβαιος ότι ε, συμφωνώ απολύτως και πολύ συχνά εξαρτάται από το, τη διαθεσιμότητα χερσαίων μεταφορών, μεταφορών σε δρόμους. Ε, βλέποντας ε, το τι συμβαίνει τα τελευταία 20-25 χρόνια, είδαμε ότι υπάρχει διαρκής ε, αύξηση των χερσαίων μεταφορών. Βεβαίως, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με την τάση αυτή και επομένως πραγματικά θα πρέπει να δούμε από κοντά το θέμα αυτό. Όσον αφορά όμως την ίδια διατροπικότητα, έτσι όπως αναφέρεται εδώ, εδώ κρατάω κάποιες επιφυλάξεις. Τώρα, η δημιουργία νέων ευρωπαϊκών οργανισμών, συγκεκριμένα δε οργανισμό για την οδική ασφάλεια ή την ασφάλεια των μεταφορών. Τι να σας πω τώρα, διαρκώς βαρύνεται η γραφειοκρατία στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες κτλ. Και επομένως δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε ακόμα ένα μανιταράκι. Νομίζω ότι καλό θα ήταν αντιθέτως να ε, μειώσουμε λίγο τον αριθμό αυτών των ε, υπηρεσιών και εν πάση περιπτώσει αντί να διαβρύνουμε τη γραφειοκρατία να δούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη ε, συγκεκριμένα στον τομέα των μεταφορών έτσι ώστε να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας και όποια γραφειοκρατία υπάρχει να είναι πιο αποτελεσματική και αντί να κάνουμε πιο αποτελεσματικά, αποτελεσματική τη διοίκηση ή τη διαχείριση ε, επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο την γραφειοκρατία. Όσον αφορά τώρα τη δημιουργία ταμείου μεταφορών και εδώ θα πω το ίδιο πράγμα. Ε, ε, νομίζω ότι επανειλημμένα το Κοινοβούλιο έχει πει ότι μάλλον υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να αφήσουμε περισσότερο ε, χώρο στα κράτη, στις, ε, ε, στις περιφέρειες. Νομίζω ότι εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει επικουρικότητα. Το να δημιουργήσουμε άλλο ένα ταμείο που στην ουσία είναι πρόφαση έτσι ώστε εμείς ε, να, έχουμε, ε, να αναμειχθούμε περισσότερο στα εσωτερικά των ε, κρατών και να αναμειχθούμε περισσότερο με αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί στην αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Είτε πρόκειται για γραφειοκρατία, είτε πρόκειται για επικουρικότητα, είτε πρόκειται για δημιουργία υπηρεσιών ή ταμείων. Δεν νομίζω ότι αυτά τα δύο θέματα με βρίσκουν σύμφωνο και δεν θα δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σας. Ευχαριστώ, η κυρία Άλβαρες. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας πω το εξή. Η διαδικασία είναι η κανονική, ναι, αλλά βλέπετε εμείς είχαμε πολύ λίγο χρόνο από τη στιγμή που πήραμε τη μετάφραση του κειμένου και το θέμα θέλει μελέτη σε βάθος, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια και για τις μεταφορές στην Ευρώπη. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπορέσαμε να πάμε σε βάθος και ζητάω συγγνώμη από τον εισηγητή γι' αυτό. Εγώ κατάλαβα στην αρχή ότι το άγγραφο του εισηγητή θα ήταν μια εναλλακτική λύση σε σχέση με το έγγραφο και την πρόταση της Επιτροπής. Όμως φαντάζομαι ότι η συγκεκριτή και αυτό θέλω να το ρωτήσω, συμφωνεί τελικά με την ανάλυση της Κομισιόν και γι' αυτό δεν δίνει άλλο εναλλακτικό κείμενο. Τώρα για να μιλήσουμε για την μελλοντική πολιτική μεταφορών στην Ευρώπη, εδώ στο Κοινοβούλιο πρέπει να ξεκινήσουμε με μία ανάλυση όσον αφορά την πολιτική και τα αποτελέσματά της μέχρι τώρα, για να ξέρουμε τι κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Πιστεύω δηλαδή ότι η Επιτροπή, ο εισηγητής, θα πρέπει να φροντίσει ώστε να ξεκινήσουμε από μια ανάλυση της κατάστασης τα τελευταία έτη. Και ξεκάθαρα και ρητά να καταλήξουμε μετά στους στόχους και τις προτεραιότητές μας σε αυτούς τους στόχους. Η μεγάλη καινοτομία της έκθεσης είναι ότι καταλήγει σε πρόταση ποσοτικής έκφρασης. Στόχους που να μπορούμε να μετρήσουμε. Αυτή τη δυνατότητα πρέπει να την έχουμε, αφού προηγουμένως όμως ξέρουμε ποια είναι η σημερινή πραγματικότητα. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, ναι, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον ρόλο των μεταφορών, τον τριπλό ρόλο στον οποίο αναφέρθηκαν και άλλοι πριν από μένα. Οικονομικός είναι ο ρόλος, κοινωνικός, ε, γεωγραφικός, διότι βοηθάει την περιφέρεια. Αυτά πρέπει να υπογραμμιστούν εν μέσω μάλιστα οικονομικής κρίσης, όπως λέει και ο συγητής. Τι ρόλο μπορούν να παίξουν μεταφορές μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Και όσον αφορά τους στόχους, πιστεύω ότι η ασφάλεια αξίζει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Γιατί η ασφάλεια είναι ζωτική σημασίας. Αναφερθήκαμε και στα τελευταία γεγονότα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Ναι, γι' αυτό και πιστεύω ότι χρειάζεται χωριστό κεφάλαιο για την ασφάλεια. Και μέσα στην ασφάλεια, και το συζητήσαμε και μαζί όταν βρεθήκαμε, είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε security και safety. Ασφάλεια και σιγουριά. Διότι από τη μια μεριά έχουμε την ασφάλεια και από την άλλη την ε, ασφάλεια που έχει να κάνει με εξωτερικούς παράγοντες. Η πολιτική μεταφορών πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες, να θέτει τους κανόνες, γιατί εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Όσον αφορά την εσωτερική αγορά και τη συνοχή είναι πολύ σημαντικό μαζί με την ασφάλεια να βάλουμε και τον στόχο εδαφικής ολοκλήρωσης. Και εκεί μέσα είναι και το τμήμα που ονομάζει εσωτερική αγορά ο κύριος Γκρός. Συμφωνώ με αυτό που λέτε, ότι δηλαδή για την οικονομική Ευρώπη οι μεταφορές είναι πολύ σημαντικές και θα ενίσχυα εγώ αυτή την ιδέα της αγοράς και τις σχέσεις της με τον πολίτη λέμε όχι σύνορα, οι οικονομικές δραστηριότητες δεν έχουν σύνορα, αλλά θέλουμε κάτι περισσότερο από την μεταφορά των εμπορευμάτων και την εσωτερική αγορά. Εγώ θα μιλούσα και για τις περιφέρειες και για τις χώρες και για τον πολίτη πάνω απ' όλα. Εδαφική λοιπόν συνοχή είναι ένα στοιχείο κλειδί και ένας κατά προτεραιότητα στόχος μας. Υπάρχει μια καινοτομία. Είναι η αποτελεσματική χρήση των συνδυασμένων μεταφορών που είπε ο κύριο Γκορ. Και ο κύριο Σέιντ πριν αναφέρθηκε στι συνδυασμένε μεταφορέ και στην αποτελεσματικότητα του συνδυασμού αυτού διαφορετικών μέσων μεταφοράς. Πέρα λοιπόν από μια ισορροπία στις μεταφορέ θέλουμε τι συνδυασμένε μεταφορές και αυτή η ιδέα πρέπει να τονιστεί μαζί με την ισορροπία στις διαφορετικές μορφές μεταφορών. Θέλουμε λοιπόν μια νέα πολιτική που να λαμβάνει υπόψη και τους υδροδρόμους και τις θαλάσσιες μεταφορές κατά προτεραιότητα βέβαια πάντα η ασφάλεια, η βιωσιμότητα των μεταφορών λαμβάνοντας υπόψη την αγορά και τον άνθρωπο. Θα ήθελα να ενισχυθεί λοιπόν στην έκθεσή σας ό,τι έχει να κάνει με τους σιδηροδρόμους και τις θαλάσσιες μεταφορές. Και ολοκληρώνω με το εξή. Έχει πολύ θάρρος ο κύριος Γκρός που μιλάει για την αναγκαιότητα χρηματοδότησης ολόκληρης αυτής της νέας, ε, μεταφορά, της νέας πολιτικής μεταφορών. Νομίζω ότι αποτελεί καινοτομία επειδή μιλάτε για ειδική μεταχείριση όσον αφορά τις επενδύσεις που γίνονται στις μεταφορές, να λαμβάνονται δηλαδή ιδιαίτερα υπόψη στο πακέτο. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και από εκεί και πέρα θα υποβάλουμε και τροπολογίες προσπαθώντας να βελτιώσουμε την πρόταση του κύριου Γκρός, τον οποίο ευχαριστώ ρητά για τον τρόπο που έχει προσεγγίσει το θέμα. Ως στη εισηγήτρια θα προσπαθήσω να συνεισφέρω επικοδομητικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, τον εισηγητή, συγγνώμη, είχα μια ενδιαφέρουσα εμπειρία διότι είχα συμφωνήσει με την Κομισιόν για τα θέματα μεταφορών εναερίων και εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι οι οποίοι είναι και μετρήσιμοι και μπορούμε να καταμετρήσουμε το επίπεδο της επιτυχίας μας. Όλα αυτά είναι αξιόλογα και θετικά αλλά υπάρχουν και κάποια σημεία όπου διαφαίνονται οι ελλείψεις της αρχικής ε, πρότασης. Όταν μιλάμε για τις ε, εναέριες μεταφορές, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν ε, αναλυθεί ιδιαίτερα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, λέμε όλα πάνε καλά τώρα, απλώς στο μέλλον πρέπει να τα κάνουμε διαφορετικά. Είναι τόσο αρνητικές λοιπόν οι τωρινές συνθήκες σήμερα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι στο μέλλον αν δεν τροποποιήσουμε το γενικό πλαίσιο. Έχουμε στρέβλωση του ανταγωνισμού, έχουμε έλλειψη ισότητας ανταγωνισμού και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την ανάπτυξη των μεταφορών. Επίσης, στον τομέα των εναρίων μεταφορών που έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις εκπομπές έχουν πέντε προνόμια ότι δεν πληρώνουν για την ε, φορολογία κυροζήνης που είναι σημαντικά ποσά έχουν ε, δώρα 85% των πιστοποιητικών εκπομπής για, την, ε, για τις εκπομπές και δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιβαρύνσεις για την πτήση πάνω, σε, πάνω από ακτικές περιοχές για την, για την Έχουμε λοιπόν αυτά τα πέντε προνόμια τα οποία απαρίθμησα σε σχέση με την αεροπορική μεταφορά. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προνόμια τα οποία είναι τεράστια. Για τους δρόμους μιλάμε για, τις, ε, ε για την ασφάλεια. Είναι πραγματικά σοβαρό το, το ατύχημα αυτό στη Χάλε μετά στους σιδηροδρόμους. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε 40.000 νεκρούς στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Αυτό είναι σημαντικό σε σχέση με τους νεκρούς από, τα, από τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν το πλαίσιο με το οποίο θα αυξήσουμε την ασφάλεια στους δρόμους. Διατροπικότητα. Ακόμα δεν ξέρω τι είναι διατροπικότητα. Αυτό είναι μια εφεύρεση της Κομισιόν. Ώστε να αντιμετωπιστεί η, η, να αντιμετωπιστεί η μετακίνηση των μεταφορών στο δρόμο. Λεγόταν προηγουμένω διατροπικότητα, τώρα λέγεται συντροπικότητα. Λοιπόν, αυτό όμως είναι μια πραγματική αντίφαση και είναι μια αντίφαση που υπάρχει μεταξύ του σημείου 3 και 4. Εμείς μας ενδιαφέρει να προωθήσουμε την αποτελεσματικότητα αλλά όταν είναι έτσι το πλαίσιο που μόνο του δρόμου μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Οδηγούμε με ένα παράλογο τρόπο στο να δίνουμε προνόμια στις οδικές μεταφορές με μια τέτοια αντιμετώπιση. Αυτά είναι λοιπόν μερικά θέματα τα οποία εγώ βλέπω να προέρχονται στο έγγραφο αυτό. Έχουμε τα στοιχεία, όπως βλέπουμε και στην έκθεση του κυρίου Γκρός, αλλά λείπει κάτι το οποίο είδα εγώ σε μία παρουσίαση PowerPoint ε, ε, στο βερίνο της ε, Κομισιόν 34% έχουν, 35% έχουν αυξηθεί οι εκπομπές για τη μεταφορά από το 1999, ενώ έχουν πέσει 10% οι εκπομπές από βιομηχανικούς κλάδους. Και είναι πραγματικά ενδιαφέρον το οποίο το λέει αυτό η Κομισιόν, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο εμεί δεν μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο. Λοιπόν, αν δεν υπάρξει μια τροποποίηση στον τρόπο μεταφορών, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και σίγουρα θα πετύχουμε το στόχο του 2020 και αυτό είναι σημαντικό. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα στις πόλεις. 70% όλων των λαβερών εκπομπών για το κλίμα προέρχονται από κινητικότητα στις πόλεις. Και βρίσκω πολύ ωραίο αυτό το οποίο λέγεται ότι πρέπει να διπλασιαστεί ο αριθμός αυτών οι οποίοι χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες. Πρέπει όμως να διπλασιάσουμε και τους ε, ποδηλάτες και τους πεζούς. Όταν βλέπουμε, Παραδείγματο χάρη σε πόλη σαν τη Ματρίτη, ότι είναι δύο μέτρα το πεζοδρόμιο και 15 μέτρα ο δρόμος, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν ευνοεί τους πεζούς προτιμάει ο κόσμος να περπατάει στον δρόμο. Ήξερα ότι αμέσως θα με, θα με αντικρούσετε. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να έχουμε μια συμπερίληψη της πτυχής του περιβάλλοντος για όλες τις μορφές μεταφορά. Η Κοπενχάγη έδειξε τι μπορεί να κάνει κανείς. Μέσα σε 10 χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 20% οι ποδηλάτες, ακόμα και στο Βερολίνο έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των ποδηλατών. Και επομένως, τα θέματα της της ηλεκτρονικής, της ηλεκτρικής μάλλον κινητικότητας, είναι τα ηλεκτρικά ποδήλατα στις πόλεις. Αλλά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα πρέπει να προωθηθούν με διάφορα κίνητρα γιατί μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τη ζημιά προς το περιβάλλον. Και τώρα το θέμα των οικονομικών αρνητικών πτυχών της, ε, των μεταφορών. Ο αυτοκινητόδρομος, ο δακτύλιος του Μονάχου κατέστρεψε πάνω από 100 μικρές ζηθοποιίες στην περιοχή αυτή. Χάθηκαν θέσεις εργασίας. Αυξήθηκε η χρήση των μεταφορικών μέσων. Λοιπόν, δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για τα πλεονεκτήματα, πρέπει να μιλάμε για την κατάργηση θέσεων εργασία, την κατάρρευση τη ποιότητα ζωή και το γεγονό ότι καταδαπανάται ένα μεγάλο μέρο του χώρου από τι υποδομέ μεταφορών. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω, κύριε Πρόβλημα. Πρόεδρε. Thank you, uh, Michael. I never realized... Michael. Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν τόσο σοβαρό αυτό το θέμα με όλε αυτέ τις ηθοποιίες που έκλεισαν. Σοβαρό πλήγμα η κυρία Γιάννα Σέντερ. Ευχαριστώ. Είναι γεγονό. Στο Βερολίνο μου φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο, στενή, πιο στενά τα πεζοδρόμια. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η πόλη. Πιο στενά από την Μαδρίτη. Εντάξει, αυτό με τα ποδήλατα με τα ελάχιστα χρήματα τα οποία έχουμε καταφέραμε να ευνοήσουμε ιδιαίτερα τη χρήση των ποδηλάτων στη Μαδρίτη. Θέλω να ευχαριστήσω τώρα ιδιαίτερα τον κύριο Γκρός και την κυρία Άλβαρες η οποία είναι σκιώδης μας εισηγήτρια για την προσπάθεια που κάνουν στο να αναπτυχθεί ένας διάλογος ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή και καινοτόμα ε, αντιμετώπιση στην έκθεση αυτή για το μέλλον των μεταφορών. Εγώ συμφωνώ με τις δύο κύριες ιδέες που έχουν τεθεί, το θέμα δηλαδή της ε, εφαρμογής να εξασφαλίσουμε ότι λειτουργεί σωστά η αγορά, ότι λειτουργούν σωστά οι μεταφορές. Αυτό απαιτεί μια σωστή εφαρμογή λοιπόν. Απλώς θα ήθελα να θέσω ορισμένες προτάσεις εδώ για να έχουμε μια αποτελεσματική διατροπικότητα θα ήταν χρήσιμο να κινηθούμε προς τους στόχους μας με ένα πιο προσεκτικό τρόπο. Νομίζω ότι αυτό θέλει να κάνει και ο κύριος Γκρός προωθώντας την αποτελεσματική διατροπικότητα. Θα ήταν όμως πιο σημαντικό να μπορέσουμε να δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτή η διατροπικότητα. Άλλο είναι τα στοιχεία των μεταφορών, της μετατόπισης από μία μορφή μεταφορά σε μια άλλη και το άλλο να δούμε τους κόμβους μέσω των οποίων μπορούν να υπάρχουν αυτές οι μετακινήσεις από ένα τρόπο μεταφοράς σε έναν άλλο. Πώς λοιπόν, πού είναι τα κομβικά σημεία στα οποία διαπλέκονται οι τρόποι μεταφορών και πώς μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Είναι σημαντικό αυτό λοιπόν να το δούμε και αυτό με οπτικό τρόπο. Και φυσικά η συμπλήρωση της εσωτερικής αγοράς εδώ δεν ξέρω αν πέραν από τις κατεχώρησιν πράξεις, η συνθήκη της Λισαβόνας έχει και νέα μέτρα για να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μέσα στα χρονικά πλαίσια που θέλουμε και με τον τρόπο που θέλουμε την εφαρμογή αυτών των ε, μέτρων. Βλέπουμε τι γίνεται με τον Γαλιλαίο, βλέπουμε τι γίνεται με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Διότι εφόσον η συνθήκη αποδέχεται μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν δεν έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό πνεύμα ώστε να εφαρμοστεί αυτό το κοινό πνεύμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει η ίδια πολιτική θέληση, αυτό είναι μια από τις αδυναμίες μας, η ίδια πολιτική θέληση για την εκπόνηση, για την εκτέλεση όλων αυτών των ε, Πιστεύω και εγώ ότι θα ήταν χρήσιμο ένα αποκεντρωμένο φορέα για τι οδικέ μεταφορέ, αλλά θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και στον τομέα των πόλεων, όπου χρησιμοποιούνται πάρα πολύ οι δρόμοι και η οδική μεταφορά. Κάπω θα πρέπει να το ενσωματώσουμε στη σύνολη αυτή προβληματική. Δεν πρέπει να χάσουμε λοιπόν το στοιχείο αυτό του αστικού χώρου που το είχαμε τονίσει στην προηγούμενη θητεία μας ποσοτικοποιημένοι στόχοι και εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε και περισσότερα στοιχεία, όχι μόνο τα λεωφορεία και τα, τα πούλμαν και τα σιδηρόδρομοι, αλλά και τα τραμ, τα οποία πρέπει να έχουν μία παρουσία στον αστικό χώρο. Για τα δίκτυα, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και φυσικά υποστηρίζω την πρόταση της κυρίας Αλβάρες για τον χρυσού κανόνα. Αεροδρόμια. Και εκεί θα πρέπει να, τους, περιλάβουμε την πρόβλημα των αεροδρομίων και σε ό,τι αφορά τους καταμετρήσιμους στόχους, το η μείωση 20% στον αριθμό των νεκρών στις μεταφορές γιατί να μην διατηρήσουμε το στόχο του 50% γιατί υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία έχουν έρθει λίγο πιο αργά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να έχουν πιο πολύ χρόνο για να επιτύχουμε το στόχο του 50% το 2010. Εγώ θα διατηρούσα το 50% σε ό,τι αφορά τα θύματα και το 40% για τους σοβαρά τραυματισμένους. Αυτό θα ήταν λοιπόν μια μεγάλη πρόκληση για τα παλιά κράτη-μέλη που έχουμε καταφέρει να μειώσουμε στο ίμι τον αριθμό των θανάτων. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα δώσουμε καλό μήνυμα πολιτικό στα νέα κρατημέλη αν περάσουμε αμέσως από το 50% στο 40%. Τέλος, οι ιδρυοδρομικές μεταφορές. Λέτε, ίσως είναι λάθος μετάφραση, ότι από το 2011 ότι θα πρέπει να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι θα, σιδηρόδρομοι θα κινούνται πια με δίζελ. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι θετικό. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό πρόβλημα ε, μετάφρασης. Τέλος, οι διατροπικές ε, πλατφόρμες όπου αναφέρεστε στα προβλήματα των ε, εσωτερικών υδατήριων δρόμων. Δεν είναι μόνο αυτό το οποίο πρέπει να υποστηρίξουμε, πρέπει γενικά να υποστηρίξουμε τι διατροπικέ πλατφόρμε και στην, ε, στα σημεία σύζευξη άλλων τρόπων μεταφορά. Κύριε Φώστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω υπερβολικά. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρόσο για αυτήν την ε, πολύ ολοκληρωμένη έκθεση, η οποία είναι πολύ ε, λογική και πρόκειται για ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην, ε, στην καρδιά του Κοινοβουλίου για πολλά χρόνια. Ο κύριος Βαντάλεν έθιξε ήδη κάποια θέματα με τα οποία συμφωνώ, δηλαδή Πιστεύω ότι σαν γενικό ε, κανόνα αυτό που θα πρέπει να προσδοκούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ξεχνάμε συχνά ε, είναι να μην είμαστε εξαιρετικά ε, περιγραφικοί μην... γιατί ξέρετε δεν νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε στοιχεία τα οποία να αποτελούν πανάκια για κάποια θέματα γιατί να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν εθνικές ιδιαιτερότητες, υπάρχουν περιφερειακές ιδιαιτερότητες, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Επίσης πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κάνει καλά και πολύ καλά πρέπει να συνεχίσει να τα, να τα κάνει. Από την άλλη πλευρά όμω υπάρχουν εθνικέ κυβερνήσει, περιφερειακέ κυβερνήσει, ενδεχομένω και κάποιες, κάποια μεμονωμένα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, ενδεχομένω ακόμα και κάποιε μεμονωμένε ε, ε, πιέσει ε, και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν αρμοδιότητες οι οποίες θα πρέπει να, ε, να ασκούνται. Ε, και κάτι άλλο, το οποίο έθιξε και ο κύριος Βαντάλ και συμφωνώ με την παρατήρησή του. Αναφέρεται ο εισηγητής σε δημιουργία ταμείου. Ωραία πολύ καλά ένα ταμείο, αλλά με τι χρήματα, από πού θα έρχονται τα χρήματα αυτά. Ε, δηλαδή μπορούμε να πούμε πολλά για ένα ε, ταμείο. Βεβαίω, διαρκώς ε, γίνεται λόγος για προτάσεις περικοπών, γίνεται λόγος για υπερβολική γραφειοκρατία. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς θα έχει προστιθέμενη αξία αυτό το, το ταμείο αν ε, ε, νομίζω ότι το να βάλουμε μέσα στο ίδιο σακί και την ανάπτυξη και την καινοτομία και την έρευνα δεν ε, μπορώ να συμφωνήσω με όλα αυτά. Απ' την άλλη πλευρά ε, όλοι αναγνωρίζουμε την σημασία ε, της, των διασυνοριακών επαφών. Μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι αποκομμένο γιατί είναι νησί, αλλά οι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκής Ένωση βεβαίω χρειάζονται πάρα πολύ καλή συνεργασία όσον αφορά αυτά τα διασυνοριακά περάσματα. Δεν δίδεται όμως αρκετή τι σημασία στην διεθνή διάσταση. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Ε, το έχουμε κάνει ήδη και με τους πράσινους για αρκετά θέματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω ότι εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρότι είμαστε νησί, έχουμε απελευθερώσει την ε, αεροπορία. Ε, και ε, νομίζω ότι ε, πρέπει να το δούμε το θέμα αυτό από κοντά γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες ε, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα προσβάσιμες. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπογραμμιστεί ακόμα περισσότερο η σημασία του θέματος αυτού. Θα πρέπει να δουλέψουμε στον τομέα της αεροπορίας και ενδεχομένως να φτάσουμε σε κάποιες, σε, σε κάποιες διατάξεις οι οποίες θα αναγνωρίζουν ότι εδώ εδώ βρισκόμαστε σε μια ολοκληρωμένη εμπορική οντότητα και επομένως θα πρέπει ε, όλα τα στοιχεία να συνάδουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, ε, επίσης, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή η συνεργασία που έχουμε με τη Γενική Διεύθυνση ε, Μεταφορών. Πολλές φορές έχουμε διαφωνήσει και πολύ καλά κάναμε και διαφωνήσαμε. Αλλά με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος η σχέση μας δεν είναι καλή. Δηλαδή δεν μπορούν να κατανοήσουν μερικές φορές ότι οι μεταφορές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ότι είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων, ότι είναι χώρος δημιουργίας εργασίας και ότι ε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της πολιτικής όλων των χωρών. Κοιτάξτε, μερικές φορές ε, σε θέματα τα οποία με απασχολούσαν, μιλώντας με κόσμο από την Επιτροπή, συγγνώμη, από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, είχα την εντύπωση ότι είναι από άλλο πλανήτη. Το θέμα δεν είναι να ε, ε, ε ναι σε κάποια στοιχεία και όχι, να ευνοήσουν κάποιους και να μην ευνοήσουν κάποιους άλλους. Είναι να κατανοήσουν συνολικά περί τίνος πρόκειται και να καταλάβουμε ότι εμείς δεν είμαστε ο καθένας στη γωνία του, αλλά είμαστε μέσα σε μια ε, ολοκληρωμένη. Ε, τι είπατε, ότι η Γενική Διεύθυνση ε, Περιβάλλοντος είναι από άλλο πλανήτη. Κύριο Κάντσια, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον συνάδελφο Γκρός για την εξαιρετική έκθεση που έχει υποβάλει. Θα ήθελα όμως να κάνω δύο-τρεις επιπλέον θεωρήσεις διάβασα το έγγραφο της Επιτροπής για τη στρατηγική του 2020 και δεν βλέπω εκεί την αηφόρο ανάπτυξη των μεταφορών. Νομίζω ότι αυτό το σημαντικό έγγραφο θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη την λειτουργία ε, των ε, μεταφορών γιατί αναπτύσσεται και η βιομηχανία και το εμπόριο μέσω των ε, μεταφορών και επομένως οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει λόγος και αναφορά στο έγγραφο αυτό. Επίσης Πρέπει να πω ότι έλειψα για λίγο γιατί είχαμε ψηφοφορία στην Ήτρε και πρέπει να σας πω ότι ψηφίστηκε ομόφωνα η έκθεσή μου ακριβώς που εισχολείται με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους ε, για το 2020 ε, και καλό μάλιστα την Επιτροπή μας εδώ να ενστερνιστεί όλα τα στην έκθεση αυτή περιεχόμενα ε, και επίσης τα όσα αναφέρονται για το σύστημα έξυπνων μεταφορών. Θα ήθελα να θίξω τώρα και το θέμα του προγραμματισμού και της πραγματοποίησης, της υλοποίησης. Ο προγραμματισμός είναι ιστορική στιγμή, ιστορικό στοιχείο και πρέπει βεβαίως να προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε τον προγραμματισμό αυτό έτσι ώστε οι ροές να μην περιλαμβάνουν μονάχα με μεμονωμένες ε, μεταφορές ή με μονομένα είδη μεταφορών αλλά να έχουν μια γενικότερη αξία ε, συμπερίληψης όλων των τρόπων ε, μεταφοράς και βεβαίως να δώσουμε σημασία στους κόμβους, στα hubs έτσι ώστε να υπάρξει πραγματική διατροπικότητα γιατί αυτό είναι το σημαντικό σημαντικότερο σκέλος της, πραγμα... της... Ε, του προγραμματισμού. Εάν καταφέρουμε τις ροές ε, των ε, μεταφορών να τις, διασυνδέσουμε συγγνώμη, σωστά με τους κόμβους, με τα hubs, τότε θα καταλήξουμε σε μια ορθή οργάνωση μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα διαχωρίζεται από τις πανευρωπαϊκές ε, μεταφορές ε, και βεβαίως θα ε, καταφέρουμε τελικά να διασυνδέσουμε αυτά τα δύο συστήματα μεταφορών γιατί θα υπάρξει η πραγματική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όσον αφορά τις μεταφορές. Δεύτερο σκέλος, η υλοποίηση. Πιστεύω ότι και ο Ισπανός Υπουργός και ο νέος Επίτροπος το επανέλαβαν και επομένως νομίζω πως είναι όριμη η χρόνη έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτό το ταμείο που αναφέρει ο Στέφος Γκρόσο στο, ε, στην έκθεσή του ε, που θα πρόκειται για ένα ταμείο που δεν θα προέρχεται απλώς από πόρους των κρατών ή της ε, Κομισιόν αλλά θα είναι κάτι πολύ ειδικό θα περιλαμβάνει μόνο θέματα ε, μεταφορών, να μην ε, απλώνεται σε ενέργεια ή σε άλλα θέματα αλλά ε, θα προσπαθεί να βελτιώσει τα μεμονωμένα προγράμματα μεταφορών ε, στις διάφορες χώρες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί αυτά που εμείς συζητούμε και προγραμματίζουμε επί σειρά ετών πρέπει να υλοποιηθούν κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σουγιάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε συγχαίρω και τον εισηγητή και τους σκιώδης εισηγητές για την εξαίρετη εργασία την οποία έκαναν και που είναι τροφή προσκέψη. Θα ήθελα να παρέμβω επί δύο θεμάτων. Πρώτον, για το Ταμείο και δεύτερον για τις ε, ε, πλατφόρμες αυτές ε, τις διατροπικές διασυνδέσεις όσον αφορά το Ταμείο. Θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή να, να προσθέσει στις παραμέτρους οπωσδήποτε την παράμετρο της ασφάλειας. Γιατί πιστεύω ότι είναι θεμελιώδου σημασία έτσι ώστε να υπάρξει σωστός διαχωρισμός των τρόπων με τον οποίο θα ε, παρέμβει το Ταμείο. Δεύτερον, πιστεύω ότι θα πρέπει να εντεχθεί και ένα κριτήριο απόδοσης ε, των ε, ε, κονδυλίων που θα χωρίζεται σε δύο φάσεις. Μία φάση λοιπόν πρώτη όπου θα δίνονται κονδύλια έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα εγγενή προβλήματα οποιοδήποτε τρόπου μεταφοράς και εξηγούμε εάν τώρα εμείς ε, προσπαθήσουμε να επιβραβεύσουμε με επιπλέον κονδύλια συστήματα μεταφορών υψηλών παραμέτρων, τότε θα δημιουργήσουμε μια εσωτερική ε, περαιτέρω διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που δεν μπορούν ακόμα να εφαρμόσουν ή δεν, ε, δεν διαθέτουν τις παραμέτρους αυτές είτε γιατί εντάχθηκαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε γιατί παρουσιάζουν έντονη περιφερικότητα και ε, επομένως ε, ε, δεν είχαν τον χρόνο έτσι ώστε να απαλύνουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την περιφερικότητα αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ε, υπάρξει εσωτερική αλληλεγγύη και μονάχα σε αργότερα σε μια δεύτερη φάση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά προς επιβράβευση των δικτύων που επιτυγχάνουν, έχουν ήδη επιτύχει τους στόχους. Γιατί εάν δεν ενταχθεί αυτή η διαφοροποίηση θα εξακολουθήσουμε να έχουμε ε, διαρκώς μία ε, Ευρώπη δύο ταχυτήτων και μάλιστα ε, η χαμηλή ταχύτητα να πηγαίνει διαρκώς και πιο πίσω. Δεύτερο θέμα, οι πλατφόρμες, αυτές οι διατροπικές διασυνδέσεις. Επ' αυτού πιστεύω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα ε, ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την εσωτερική ναυσιπλοεία. να ε, ε, υπάρξει η έννοια εσωτερικής λεκάνης Πλοίας, ε, που θα πρέπει να θεωρηθεί σαν σύστημα εσωτερικών ε, ε, οδών, εθνικών εσωτερικών πλωτών οδών. Δηλαδή, στην ουσία λέω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε ένα σύστημα σαν αυτό που υπάρχει ανάμεσα στα ελληνικά νησιά, θαλάσσιες διαδρομές ε, όπως αυτές λοιπόν των ελληνικών νησιών, ένα είδος τέτοιου είδους, ε, ένα είδος τέτοιου δικτύου το οποίο ε, θα αφορά όμως τις εσωτερικές πλωτές οδούς θα ήθελα να παρακαλέσω τον εισηγητή να προωθήσει ε, αυτήν την ε, ιδέα στο εσωτερικό της έκθεσης του. Ευχαριστώ πολύ ε, και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Γιάνγκ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστώ και τον κύριο Γκρός για τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και την κυρία <laughs> Φώστερ για την γενική μας διεύθυνση να πω κάτι για την έκθεση. Προφανώ εμεί θα αναμείνουμε το τελικό κείμενο της έκθεσης και την συλλογική σοφία της Επιτροπής σα, Αλλά θέλω παρόλα αυτά να μοιραστώ μαζί σα μερικά προκατακτικά σχόλια. Η Κομισιόν χαιρετίζει την έκθεση αυτή, η οποία υποστηρίζει τι κύριε πολιτικέ κατευθύνσεις του Προέδρου Μπαρόσο για την μείωση της χρήσης άνθρακος, τη λεγόμενη απανθρακοποίηση, και επίσης του Επιτρόπου κυρίου Κάλλας. Χαιρετίζουμε επίσης και τους στόχους οι οποίοι διατυπούνται σε αυτή την έκθεση, ιδίω για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πιο αποτελεσματική διατροπικότητα για μια κοινή αγορά του σιδηροδρόμους και στις οδικές μεταφορές, για μια εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και φυσικά θέλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο μέσω χρηματοδότησης των μεταφορών. Σε ό,τι αφορά την καταμέτρηση των στόχων, εσείς αναφερθήκατε στο 2020 και όχι στο 2010. Νομίζουμε ότι παρισέφρισε ο δαίμον του τυπογραφείου στα συμπεράσματά σας. Εάν όχι, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι όλοι στόχοι κακοί. Δεν μπορείτε να κάνετε λάθος όταν ζητάτε ένα εθελοντικό στόχο για τη μείωση των θανάτων στο δρόμο. <clears throat> Αλλά οι προτάσεις σας, όπως ε, τη μια φορά, δημιουργία ενός νέου ε, αποκεντρωμένου φορέα για την οδική ασφάλεια, προσκρούν ίσω την επικουρικότητα. Και νομίζουμε ότι χρειάζονται επίσης και κάποιες ε, περαιτέρω θεωρήσεις όταν μιλάτε για ποσοτικοποιημένους στόχους. 20% στη μείωση των θανάτων στον δρόμο αυτός είναι ένας ειδικό τομέας, αλλά θα έπρεπε να δούμε και την αλληλεπίδραση με την επίτευξη των στόχων διοξιδίου του άνθρακος σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά και την ανανεώσιμη, τις ανανεώσιμες μορφές μεταφορών. Επίσης, η μείωση της χρήσης ηλεκτρισμού θα απαιτούσε περαιτέρω ανάλυση γιατί δεν νομίζουμε ότι θα μείωνε συνολικά τις εκπομπές από τον τομέα μεταφοράς. 20% μείωση της εκπομπής ρήπων από τα αεροπλάνα είναι υπερφιλόδοξος στόχος κατά την άποψη της Κομισιόν και εμείς θα έπρεπε να εξετάσουμε κατά πόσο υπάρχουν πιο ε, σε σχέση με το κόστος μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των εκπομπών. Αυτά είναι όλα προκατακτικά σχόλια. Θα περιμένουμε για την τελική σας έκθεση και σε στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 η Κομισιόν έχει αρχίσει να επεξεργάζεται τη νέα λευκή βίβλο και θα ξεκινήσει η εξωτερική διαβούλευση στο δεύτερο εξάμεινο του 2010 και η εννοείται ότι βασιζόμαστε σε εσά και το συλλογικό σας έργο για να επιτύχουμε μαζί τα σωστά αποτελέσματα για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Κύριε Γκρός, θέλετε να επανέλθετε να συνοψίσετε. Σας παρακαλώ σύντομα. Βεβαίως κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι όσο το τον πιο σύντομος και συνεκτικός. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προλαλήσαντες για τη συμβολή τους στη συζήτηση και αυτούς οι οποίοι δεν συμφωνούν ακόμα με τις συγκεκριμένε μου προτάσεις τουλάχιστον αυτό μου δίνει το πλεονέκτημα να ξέρω πού βρισκόμαστε που θα βρεθούμε στην επικείμενη συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω και την Κομισιόν. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή μας έχουμε κρατήσει τα θέματα μεταφορών στο κέντρο της συζήτησης και αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό. Δεν μπορούμε πάντα να έχουμε ιδιαίτερη κατανόηση για προσεγγίσεις οι οποίες θέτουν στο κέντρο των μεταφορών ζητήματα όπως το περιβάλλον. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα στον τομέα μεταφορών. Εκεί βρίσκεται και η εμπειρογνωμοσύνη που μπορεί να προσφέρει η Επιτροπή μας στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθε. Δεν μπορώ τώρα να διεξέλθω όλες τις μεμονωμένες παρατηρήσεις θα σταθώ σε ορισμένα σημεία, κυρία Φώστερ, πραγματικά είναι σαφές ότι οι δύο πτυχές του αποκεντρωμένου φορέα που προτείνεται και του Ταμείου για τις μεταφορές φαίνεται ότι είναι προβληματικά. Άλλοι συνάδελφοι υποστήριξαν την θέση μου. Εγώ φυσικά είμαι έτοιμος να συζητήσω μαζί σας. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χρηματοδοτικό μέσο, αυτό το μέσο θα πρέπει να εξασφαλίσει και κάποια αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να δίνει να έχει κάποια κίνητρα για να λειτουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προφανώς θα είναι κάτι το οποίο θα είναι συμπληρωματικό της εθνικής ή περιφερειακής πολιτικής. Δεν πρόκειται να την υποκαταστήσει. Είναι χρήσιμο και για την αξιοπιστία μας αν όλα αυτά τα οποία υποστηρίζουμε σε θεωρητικό επίπεδο αντανακλώνται και στη δράση μας για τον αποκεντρωμένο φορέα. Εγώ υποστηρίζω τους φορείς οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί και έχουν ένα ευρωπαϊκό ρόλο. Πιστεύω ότι τα θέματα της οδικής ασφάλειας είναι τέτοια θέματα που πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι εάν εμείς αύριο θέλουμε να έχουμε ένα, μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, σε πολλούς τομείς συμβαίνει αυτό και διαπιστώνουμε ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν λειτουργούν με συνεκτικό τρόπο και δεν προωθούν ένα ευρωπαϊκό τρόπο ρύθμισης, τότε πιστεύω θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο των αποκεντρωμένων φορέων και να τους ενισχύσουμε σε συνεργασία με την Κομισιόν σε ό,τι αφορά τώρα την ενιαία αγορά. Και εγώ είμαι από αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι η εσωτερική αγορά είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα σημαντικό στόχος το να ολοκληρώσουμε την ενιαία αγορά. Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος του περιβάλλοντος και του κοινωνικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό τονίζω και εγώ στο κείμενο. Κύριε Κράμερ, οι αρνητικές επιπτώσεις. θα σας ε, δώσω τη δυνατότητα και σήμερα ακόμα να μου δώσετε τα στοιχεία αυτά και δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα, τα, τα αριθμητικά στοιχεία να τα περιλάβω στην έκθεσή μου. Μπορούμε να θέσουμε και περαιτέρω ιδέες και αυτό αφορά ιδιαίτερα για τα ποσοστά τα οποία αναφέρατε. Αναφερθήκατε στην ασφάλεια στις ενέργειες μεταφορές και στις ε, οδικές μεταφορές. Αλλά αυτά είναι απλώς στοιχεία τα οποία έχουν ε, αναφέρει οι εμπειρογνώμονες. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικά τους θανάτους και αυτή τη στιγμή ο στόχος μας είναι έχοντας κατέβει στο 60% των θανάτων σε σχέση με πριν από 10 χρόνια θέλουμε να κατέβουμε άλλα 40%. Επομένως αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα στόχο να μειώσουμε κατά 80% τους θανάτους σε σχέση με την κατάσταση πριν από 10-15 χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θυματικό. Έχουμε την ίδια αντιμετώπιση λοιπόν κύριε Κράμερ. Κύριε Ελχαντραουή, εγώ γνωρίζω ότι το ατύχημα στο Βέλιο, το σιδηροδρομικό ατύχημα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει σε καλύτερη στοχοθεσία Στι ε, συνδρομικέ μεταφορές και το έχω αναφέρει αυτό στην ε, έκθεσή μου. Έχουμε τις τεχνολογίες που χρειάζονται για την ασφάλεια. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν την καλύτερη δυνατή τεχνολογία. Και εγώ γι' αυτό αναφέρω στην εκθεσή μου όλα αυτά τα οποία γίνονται, οι τεχνολογικές αυτές εξελίξεις να είναι τουλάχιστον διαλειτουργικές. Δεν έχει νόημα λοιπόν να φτιάχνουμε νέες υποδομές οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες διαθέσιμες τεχνολογίες και δεν προωθούν την διαλειτουργικότητα με άλλες ε, υποδομές. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια τέτοια δράση που θα επιτρέψει και θα επιβάλλει ενδεχομένω να υπάρχει αυτή η διαλειτουργικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν για όλα αυτά που είπε η φιλελεύθερη ομάδα για την ε, εσωτερική αγορά. Νομίζω ότι η ολοκλήρωση τη εσωτερική αγορά, όπω είπα προηγουμένω, είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε την ολοκλήρωση τη εσωτερική αγορά με οτιδήποτε τίμημα. Έχω δώσει, ελπίζω, και μια απάντηση στου πράσινου και εν τέλει, σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Κάσιαν, <clears throat> ότι εάν δεν είναι αρκετά ισχυρή η διατύπωσή μου για την ε, αηφόρο ανάπτυξη στον τομέα των μεταφορών, επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είπα, ότι δεν πρέπει να δούμε τις μεταφορές μονάχα ως ένα ζήτημα του περιβάλλοντος, αλλά ως ένα στοιχείο οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν το ρόλο των μεταφορών και πιστεύω ότι και ο αρμόδιος επίτροπος θα υποστηρίξει ιδιαίτερα αυτή την πτυχή των μεταφορών. Και κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μην είναι πολύ μακρύ το χρονικό πλαίσιο για τις τροπολογίες, αλλά να έχουμε αρκετό καιρό για να κάνουμε τη συζήτηση των τροπολογιών μεταξύ μας, ώστε στη συνέχεια επί τη βάση των προτάσεων των συναδέλφων, μέσα στις ε, επόμενες τρεις εβδομάδες, να μπορούμε να έχουμε λοιπόν επί τη βάση αυτών των προτάσεων τη συζήτηση το Μάρτιο και ιδίω να μπορέσω να συζητήσω με τους σκιώδεις συγητέ και τους άλλους ενδιαφερόμενους για να προχωρήσουμε σε ένα εντατικό διάλογο κάτι το οποίο θα διευκολύνει και την εξέταση των τροπολογιών και την ψηφοφορία τους. Επομένως, θα μπορούσαμε να έχουμε <clears throat> ένα μήνα για την κατάθεση τροπολογιών και μέσα σε έξι εβδομάδες να μπορέσει να υπάρξει συζήτηση για αυτές τις τροπολογίες ώστε η τελική ψηφοφορία θα μπορούσε να είναι τον Απρίλιο ή το αργότερο τον Μάιο ώστε το έγγραφο αυτό να μπορεί να μπορέσει να έρθει στην Ολομέλεια πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ευχαριστούμε. Κύριε Γκρός. Για την προθεσμία τροπολογιών είχαμε πει 1η Μαρτίου. Αν θέλετε να το παρατείνουμε, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά τότε το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για τους άλλους τομείς. Συστήνεται λοιπόν μετά την 1η Μαρτίου. Εντάξει. Αλλά τότε πρέπει κι άλλα να αλλάξουν. Σας προτείνω τρεις ή τέσσερις εβδομάδες τουλάχιστον να αφήσουμε ώστε να ακούσουμε τις προτάσεις από όλους τους συναδέλφους και να κατατεθούν υπομορφή τροπολογιών. Τότε προτείνω να πούμε 15 Μαρτίου. Τότε έχουμε τέσσερις εβδομάδες. Και δεν μπερδευόμαστε και με το Πάσχα. Έτσι. 15 Μαρτίου λοιπόν προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών και βέβαια πρέπει να δούμε το χρονοδιάγραμμα για μετά. Ινές. Αυτό σημαίνει ότι θα ψηφίσουμε τον Μάιο στην Επιτροπή ή στην Ολομέλεια. Στην Ολομέλεια. Για να προλάβουμε το Συμβούλιο του Ιουνίου. Νομίζω ότι είναι στην Ολομέλεια. Θα προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε τον Μάιο. Αλλά πρέπει να το δούμε ακόμα. Καλά τα λες, αλλά αν αποφασίσουμε να αναβάλουμε την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, εννοείται ότι πρέπει να δούμε μετά πότε θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας, ανάλογα με τις ημερομηνίες συνεδριάσεως της Επιτροπής μας και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Καταρχήν λέμε 15 Μαρτίου προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Εντάξει. 15 Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Κατοχυρώθηκε. Ωραία, σας ευχαριστώ. Τώρα βέβαια έχει περάσει ο χρόνος. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να ε, κερδίσουμε χρόνο. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Έκθεση του κυρίου Λάχφριντ. Έχουμε 80 τροπολογίες, αλλά φαίνεται ότι βολεύονται κάπως. Τέλος πάντων, για να δω, ο συμφωνεί μαζί μου γι' αυτό. Κύριε Λάιτφρυντ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσω και εγώ να κερδίσω λιγάκι χρόνο και να μην μακρηγορήσω. Αν θέλετε να είμαι συνοπτικός, να συνοψίσω. Νομίζω ότι υπήρξε μεγάλη συμφωνία μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και του εισηγητή για τα θέματα αυτά των τελών ασφαλείας. Έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Πρόεδρε στο ότι πολλές από τις τροπολογίες επικαλύπτονται ή και ταυτίζονται κιόλας και αυτό ίσως οφείλεται σε μια αποτελεσματική άσκηση πίεσης από τα λόμπι. Πάντως, ο στόχος μας είναι στο τέλος να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και να κάνουμε στο δυνατόν πιο αρμονική και γαλήνια την ε, ψηφοφορία. Μία από τις κατευθύνσεις στις οποίες <clears throat> απευθύνονται οι τροπολογίες ζητά να ληφθούν υπόψη τα δίκτυα των αερολιμένων. Εδώ όμως πολλές φορές υπάρχει η ψευδέστηση, η λαθασμένη εντύπωση μάλλον ότι εγώ δεν έχω λάβει υπόψη αυτό το θέμα. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες οι οποίες προτείνουν μια διαφορετική διατύπωση για να ρυθμιστεί το θέμα αυτό των δικτύων αερολιμένων. Επίσης συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό <clears throat> για το θέμα του πώς μπορούν να πληροφορηθούν οι επιβάτες για τα μέτρα ασφαλείας και την ε, αποζημίωση για τα μέτρα αυτά ασφαλείας. Καταρχήν, ένας τρόπος είναι να εκπροσωπούνται οι ενώσεις των καταναλωτών στα, στους φορείς όπου γίνεται η συζήτηση για τα μέτρα αυτά και όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι είναι χρήσιμο να μπορούν να παρέχονται πληροφορίες σε σχέση με τα θέματα ασφαλείας και τα τέλη ασφαλείας. Βέβαια, αυτό δεν δημιουργεί αυτομάτως μια δημοκρατική δυνατότητα συμμετοχής. Καταλήγουμε, καταλήξαμε σε μια ε, συμβαστική λύση να ληφθούν υπόψη και οι δύο δυνατότητες σε αυτή την περίπτωση και της συμμετοχής και της απλής πληροφόρησης. Για τους ε, πράσινους έχουν θέσει κάποιες τροπολογίες που δεν είναι τεχνικού χαρακτήρα, είναι εξόχως πολιτικές ε, τροπολογίες που για μένα είναι πολύ σημαντικές και υποστηρίζω αυτό το οποίο ζητούν. Οι μόνες τώρα διαφορές απόψεων μεταξύ μας περιορίζονται σχεδόν αποκλειστικά στο επίπεδο στο μέγεθος των αερολιμένων που θα πρέπει να απελαμβάνονται σε αυτό το, στην αυτού του νομοθετήματος. Υπάρχουν τρεις απόψεις. Άλλοι λένε να είναι όλοι οι εμπορικοί αερολιμένε. Μια δεύτερη προσέγγιση ορισμένων που έθεσαν τροπολογίες είναι να προσπαθήσουν <clears throat> να έχουν μόνο τους εμπορικούς αερολιμένες πάνω από ένα εκατομμύριο επιβάτες το χρόνο και η άλλη, η τρίτη άποψη είναι πάνω από 5 εκατομμύρια ε, επιβάτες το χρόνο. Είναι θέμα γούστου κατά κάποιο τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια τέτοια διαφοροποίηση σε σχέση με, με το μέγεθος του αρολιμένα, αλλά σε θέματα ασφάλειας εγώ νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο να διαφοροποιήσει κανείς το επίπεδο ασφάλειας ανάλογα με τον αριθμό των επιβατών. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες οι οποίες αφορούν μια δυνατότητα καθυστέρησης εφαρμογής αυτών των τελών ασφαλείας. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι αυτό έχει νόημα να γίνει κάποια τέτοια καθυστέρηση τη στιγμή που έχουμε όλοι αποδεχτεί να υπάρχουν αυτά τα τέλη ασφαλείας τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο κόστος των ε, αεροπορικών μεταφορών. Νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία να έχουμε εφαρμογή των λεγόμενων πιο αυστηρών μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν για την ασφάλεια σε αεροπορικές κινήσεις. Τώρα, πώς μπορεί αυτό να είναι συμβατό με μηχανισμούς που θα οδηγήσουν σε καθυστέρηση της επιβολής των τελών, δεν είναι σαφές. Δεν έχει πολύ νόημα κατά τη δική μου άποψη. Και εξάλλου, εκτός από την ε, τροπολογία των ε, φιλελευθέρων την 87 ε, εκεί έχω ένα πρόβλημα γιατί ήταν στα αγγλικά και περίμενα από την κυρία Πλάσερτ να μου κάνει μια καλύτερη διευκρίνηση για το τι ακριβώς θέλει η φιλελεύθερη εκεί. Εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την πολύ καλά καμωμένη έκθεση. Και είμαι ιδιαίτερο ευτυχής που καταφέραμε να φτάσουμε σε συμβιβαστικές λύσεις σε πολλά σημαντικά θέματα πρέπει να πω ότι και στις επόμενες μέρες είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε και το θέμα της διαφάνειας ε, όσον αφορά το κόστος το οποίο θα βαρύνει τους επιβάτες δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να επιβαρυνθούν ε, περαιτέρω. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να πληροφορηθούν το κόστος, ε, να έχουν συγκεκριμένη πληροφόρηση για το κόστος το οποίο θα πρέπει να τους επιβληθεί με την έννοια ότι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση ότι αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας. Κατά τα λοιπά δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χένες Πλασάρτ και το πρόβλημα ε, της τροπολογίας 60 ήταν κάποια άλλη εν περιπτώσει. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη και εγώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εισηγητή. Έκανε κάποιες παρατηρήσεις για τα δίκτυα αερολιμένων. Εγώ εδώ και μήνες το λέω. Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τις διαφορές που υπάρχουν. Ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Πάντως, Συμφωνώ με αυτά που λέτε για την τροπολογία των... Ε, μάλλον δεν συμφωνώ με την τροπολογία των πρασίνων. Μπορεί να είναι πολύ καλή, αλλά δεν συμφωνώ με αυτήν. Τώρα, για την τροπολογία, ποια ήταν, 66? Εδώ ήταν για τους χρήστες των αεροδρομίων όσον αφορά την ενημέρωσή τους για το κόστος της ασφάλειας και τη χρηματοδότηση που πρέπει να παρέχεται από τον φορέα που έχει την ευθύνη επιβολή τελών ασφαλείας. Πρόκειται για τους κομβικούς δείκτες επίδοσης σχετικά με την ασφάλεια. Λυπάμαι που πρέπει να φύγω όμως τώρα. Πάντως για την τροπολογία αυτή που είναι η αριθμός 67 ναι, θέλω να την υπερψηφίσετε. Τροπολογία 67 ήταν τελικά. Εντάξει, κυρία Πλασέρτ, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλά βέβαια τα πράγματα, αλλά κύριε Λίχτεμπεργκε τώρα από τους Πρασίνους, παρακαλώ. Ευχαριστώ, αγαπητέ κυρία Πρόεδρε. Εγώ βρίσκω πολύ συμπαθητικούς τους φιλελεύθερους, αλλά δεν μπορώ να υποστηρίξω προτάσεις τους, οι οποίες υποστηρίζουν ουσιαστικά το κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτό είναι το όριο της συμπαθίας μου. Δεν μπορώ να φτάσω σε αυτό το σημείο για τα σημαντικά θέματα στον τομέα αυτό. Μπορούμε να πούμε ναι στη διαφάνεια, πολύ σωστό είναι αυτό, και ιδίως στις αεροπορικές μεταφορές, όπου υπάρχουν πολλές επιδοτήσεις και ενκρυπτό επιδοτήσεις στον τομέα αυτό. Είναι απόλυτα κατεπήγον να υπάρξει διαφάνεια. Επομένως είμαι υπέρ οποιασδήποτε πρόταση η οποία προωθεί την διαφάνεια στον τομέα αυτό και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το παραμελήσουμε γιατί δεν μπορούμε να κρατάμε τα μάτια μας κλειστά. Στο θέμα της ασφαλείας θα πρέπει να είναι πολύ σαφές το σύνολο των κανόνων. Έχουμε την εμπειρία των ε, κρυφών επιδοτήσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Έχουμε λειτουργήσει στο παρελθόν με μεγάλη αδιαφάνεια, μεταφέρονται από τον ένα στο άλλο οι διάφορες πηγές κόστους <clears throat> και εγώ νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια δημόσια συζήτηση για το ζήτημα της διαφάνειας. Σε ό,τι αφορά τώρα το ποιος θα φέρει το κόστος. Εγώ δεν θεωρώ ότι να κατανοήσω γιατί θα πρέπει εμείς να είμαστε όμοιροι αυτής της πολιτικής. Γιατί θεωρώ ότι είναι για μένα τελείως λανθασμένες οι θέσεις των κρατών μελών που με το πρόσημα της διεθνής, διεθνούς τρομοκρατίας οδηγούν σε αυτή την αύξηση του κόστους των αεροπορικών μεταφορών. Και δεν μπορούμε να ζητούμε να πληρώσουν τα κράτη-μέλη ή ο καταναλωτής χωρίς να υπάρξει μια ευφυής ανάλυση κινδύνων. Αυτό φάνηκε και με το θέμα των υγρών και επίσης των σαρωτών πλήρους σώματος. Όταν πρόκειται για να αγοράσει κανείς αυτό το πολυδάπανο εξ, ε, εξοπλισμό έρχονται οι καλύτεροι εμπειρογνώμονες και λένε βέβαια όλα αυτά είναι απαραίτητα διότι τρέχει το σάλιο τους με τη δυνατότητα να λύσουν όλα αυτά τα προβλήματα σε τεχνικό επίπεδο. Αλλά όταν πρόκειται για το προσωπικό το οποίο, το οποίο εργάζεται στα αεροδρόμια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα θέματα της δικής τους ασφάλειας. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια σωστή κατανομή του κόστους, αλλά δεν νομίζω <clears throat> ότι είναι σωστό να υπάρχει μια αυθαίρετη εφαρμογή ε, μέτρων τα οποία δημιουργούν απλώς μια ψευδέστηση ασφαλείας αλλά δεν αντιμετωπίζουν την πραγματική, τους πραγματικούς κινδύνους. Υπάρχουν πολλά προβλήματα ασφάλειας τα οποία δεν μπορούν να επιληθούν στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ της απαραίτητης ασφάλειας και των μικρών παιχνιδιών που θέλουν να παίξουν κάποια κράτη-μέλη. Για μένα το καλά, καλά εκπαιδευμένο προσωπικό στα αεροδρόμια είναι πάντα η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια στα αεροδρόμια και γι' αυτό εγώ σας ζητώ να υποστηρίξετε την τροπολογία μας. Κατά άλλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φρίντ για τις μεγάλες προσπάθειες που έχει καταβάλει για να υπάρξει πραγματικά μια συμβιβαστική και κοινά αποδεκτή λύση στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Φώστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Λάιγκφρετ γιατί ε, είχαμε μια σειρά καλών συναντήσεων και ορθών συζητήσεων. Νομίζω ότι όλοι ακολουθούμε τον, ε, την ίδια κατεύθυνση και υπάρχουν τρία πεδία επί των οποίων είχαμε κάποιες διαφορές απόψεων. Το πρώτο σημείο το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα σχετικά με τα επιπλέον μέτρα ασφάλειας. Γνωρίζουμε ότι δεν θέλει καθόλου το Συμβούλιο, απεχθάνεται την ιδέα αυτή. Α, ε, ε, πιστεύουμε, ο, πιστεύουμε, εξακολουθούμε να πιστεύουμε λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πληρώσουν για τα επιπλέον μέτρα ασφάλειας ε, τα οποία έχουν επιβάλει στη βιομηχανία της αεροπορίας ε, και στους ε, επιβάτες. Κοιτάξτε, τώρα έχουμε καινούργια ζητήματα, τα θέματα των σαρωτών. Γίνεται μεγάλος λόγος ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι λιγότερο υπέρ. Είμαι, ε, ε, δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την κατάσταση και ούτε συμφωνώ με την τροπή που παίρνει η συζήτηση. Ο εισηγητής λέει ότι συζητήσαμε το θέμα και μάλιστα συζητήσαμε λίγο τον, τον στόχο ή τον σκοπό αυτών των νέων μέτρων ασφαλείας Όσον αφορά τώρα αυτό, αυτή την οροφή των 5 εκατομμυρίων, έχω πρόβλημα με το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το άχθος και το διοικητικό αλλά και το οικονομικό. Ε, κοιτάξτε, από την άλλη πλευρά, εάν κανείς ε, ε, παίξει το χαρτί της διαφάνειας και πει ναι, μα αυτό είναι το σημαντικό θέμα και ότι ναι, καλύπτει το κόστος αλλά μέχρι 5 εκατομμύρια, τότε υπάρχει αντίφαση εδώ. Ε, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να δούμε το σύνολο των αεροδρομίων σαν οντότητες. Δεν έχει έννοια να δούμε πόσος κόσμος περνάει από το κάθε ε, αεροδρόμιο. Τι να σας πω τότε, ε, ε, τότε η κάθε χώρα να βρει ένα σύστημα το οποίο θα αφορά τα αεροδρόμια της και που δεν θα είναι εξαιρετικά μπερδεμένο και δεν θα είναι πολύ περίπλοκο και δεν θα είναι πάρα πολύ ακριβό. Όσον αφορά τώρα τους επιβάτες και μάλλον τους εκπροσώπους ομάδες επιβατών που θα, θα αναμειχθούν στην διαβούλευση. Ε, νομίζω ότι οι αρχές θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι υπόλογες ε, στους πελάτες όσον αφορά τις επιλογές και στους επιβάτες όσον αφορά ε, τις διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν. Νομίζω ότι that they're listen Νομίζω ότι όσον αφορά ε, τα μέτρα ασφάλειας, βεβαίως αυτά γίνονται τελικά για την προστασία των των επιβατών ε, και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ε, διαφάνεια αλλά τι να σας πω τώρα εάν κάθε φορά επιβαρύνεται το κόστος του εισιτηρίου, τουλάχιστον το κόστος αυτό θέλω να διαρθρώνεται σωστά, θέλω να το βλέπω, να το ξέρω και να είναι ένα λογικό και δίκαιο κόστος. Νομίζω λοιπόν ότι στο τέλος ε, φτάσαμε σε ένα καλό συμπέρασμα με τον ε, ε, Λάικφριντ και νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον να δούμε προς τα, που θα πάει το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντουβεράκ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή κυρίως όσον αφορά τις προτάσεις του για την χρηματοδότηση της ε, ε, ασφάλειας ε, της αεροπορίας των αεροπορικών μεταφορών. Ε, εδώ και χρόνια συζητάμε ε, το θέμα αυτό και λέμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πληρώσουν για το επιπλέον βάρος και κόστος της ασφάλειας. Εδώ δεν προσπαθούμε να υπεραμυθούμε μονάχα των ε, δικαιωμάτων των επιβατών αλλά των πολιτών γενικότερα και άλλωστε την 11η Σεπτεμβρίου αυτοί που έχασαν τη ζωή τους δεν ήταν μονάχα οι επιβάτες των αεροπλάνων αλλά ήταν και απλοί πολίτες. Ε, ε, μπορούμε να δεχτούμε ότι ε, μονάχα αυτά τα μέτρα, τα επιπλέον μέτρα ασφάλειας είτε εν μέρη είτε εξ ολοκλήρου θα πρέπει να ε, χρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη και ε, αυτό, ε, γι' αυτό συμφωνώ και με την 29 του εισηγητού. Δεν πιστεύω πάντως ότι ο στόχος της οδηγίας στην ουσία της αρχικής, η αρχική ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα ασφάλειας και νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να διατηρήσουν το ισχύον σύστημα ε, καταβολής ε, των ε, τελών. Άλλωστε στην Ιταλία, στην Γαλλία και στην Ισπανία έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα, έχουν δημιουργηθεί οργανισμοί όσον αφορά την καταβολή των τελών αυτών και κατά αυτή την έννοια έχω υποβάλει την τροπολογία 79. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ρικέ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσει κανείς και το έκανε ικανοποιητικά. Ε, έχω περιέργεια όσον αφορά τις δύο τροπολογίες των πρασίνων για λόγους που μπορώ να κατανοήσω Υπάρχει η τροπολογία 37, ναι βεβαίως δεν θα πρέπει να είναι κυρωτικά προς τους επιβάτες μέτρα ασφάλειας ή μέτρα οικολογικά. Όμως αναρωτιέμαι εάν η τροπολογία αυτή δεν μπορεί να υπονοήσει ότι θα πρέπει να χαλαρώσουν τα μέτρα ασφάλειας για ε, ορισμένες ε, μορφές ε, μεταφορών. Δεν είναι ο στόχος και ο σκοπός της τροπολογίας, το καταλαβαίνω. Αλλά λέω, ενδεχομένως να υπάρξει αυτή η παρανόηση και μάλιστα εδώ κάνω και τη διασύνδεση με το σιδηρόδρομο γιατί και εκεί είχαμε τα ίδια προβλήματα ασφάλειας. Για τον σιδηρόδρομο δεν υπάρχει τέτοιου είδους μέτρο ασφάλειας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να ε, ε, πούμε, να γίνει συγκεκριμένη αναφορά στον ε, σιδηρόδρομο. Επομένως, από τη στιγμή που δεν υπάρχει τέτοιου είδους, τέτοιου είδους μέτρο, πώς είναι δυνατόν να το ενδυναμώσουμε ή να το εντείνουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε απλώς μια γενικότερη διατύπωση, δηλαδή να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στην δημοκρατία. Ε, δεύτερο, δεν έχω δεύτερη τροπολογία, δεν έχω διαβάσει το κείμενο στα γερμανικά, αλλά εν πάση πτώση λέει ότι ε, μέσω της ε, ενίσχυσης των επενδύσεων για την ασφάλεια των αεροδρομίων δεν θα πρέπει τελικά να έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων για τα αεροδρόμια. Νομίζω ότι η διατύπωση δεν είναι σωστή. Θα υπάρξουν οικονομίες καταλαβαίνουμε ποιο είναι το αρχικό πνεύμα. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνουν επενδύσεις με στόχο ε, την μείωση των θέσεων απασχόλησης, ε, των κοινωνικών και εκτιμένων δικαιωμάτων κτλ. Ε, νομίζω ότι στα γαλλικά τουλάχιστον η λέξη εφέ δεν αποδίδει το σωστό νόημα και επομένως νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε στόχο, να βάλουμε τη λέξη but στόχο και όχι εφέ αποτέλεσμα ή αντίκτυπο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το θέμα της διαφώτισης των επιβατών σε σχέση με το κόστος της ασφάλειας. Τι σημαίνει αυτό, σε τι τάξη μεγέθους βρισκόμαστε, πόσο θα κοστίζει αυτό για κάθε επιβάτη σε μία μέση πτήση. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε πόσο κοστίζει παραπάνω πραγματικά ένα σαρωτή σώματος. Δεν ξέρω λοιπόν τι θα, ποιο είναι το κόστος το, και τι αγοράζει για τον, για τον ε, επιβάτη αυτό το κόστος. Θα ήθελα η Κομισιό να μας πει ακριβώς γιατί τάξη μεγέθους κόμματο, ε, κόστους μιλάμε. Στα γερμανικά αεροδρόμια μας είπαν ότι το κόστος είναι μεταξύ 70 σεντ και ένα ευρώ και 20 και είπαν ότι αυτό θα, η εισαγωγή των σαρωτών σώματος θα προσθέτει 30 λεπτά ακόμα του ευρώ, 30 εκατοστά του ευρώ. Αλλά αυτό δεν πρέπει να το συγχαίουμε με τις ενέργειες οι οποίες θα γίνουν από τις εσωτερικές, από τις εσωτερικές αστυνομικές αρχές στα αεροδρόμια, οι οποίες ούτως ή άλλως θα ενισχύσουν τις δραστηριότητες τους. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει αν σημαίνει αυτή η αλλαγή στα αεροδρόμια ότι δίνουμε χρήματα σε, τρί, σε τρίτους, σε ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας και εκεί να ξέρουμε πόσο, ακριβώ πόσο ακριβώς θα κοστίσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει κύριε Λάκτφριντ νομίζω ότι έχετε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορεί να υπάρξει μια συνεργατική λύση που θα την υποστηρίξουν όλοι εδώ. Ευχαριστούμε κύριε Κιούν. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλω να πω και εγώ δύο λόγια. Είμαι υπέρ της τροπολογίας 29. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι οι επιβάτες πρέπει να πληρώνουν για όλα τα μέτρα ασφάλειας ε, όταν πρόκειται για τρομοκρατικές ε, επιθέσεις και ότι δεν είναι τα κράτη, οι αεροπορικές εταιρείες, οι επιβάτες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. η Lufthansa, η Air ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Αν γίνεται μια επίθεση λένε, ε, αν γίνει στη Γαλλία για παράδειγμα, η Γαλλία πρέπει να φροντίσει να τις αποφύγει. Εδώ υπάρχει μια ανομαλία δηλαδή. Όταν έχουμε να κάνουμε με την ασφάλεια, άλλοι τομεί για τους για άλλου τομεί ε, πληρώνει το κράτο. Όταν πρόκειται για τι αεροπορικέ μεταφορέ, όχι, πρέπει να πληρώνουν οι επιβάτε. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και στηρίζω απόλυτα την τροπολογία 29. Το είπαν και άλλοι στη συζήτηση. Το Συμβούλιο θα το καταπολεμήσει με νύχια και δόντια. Αλλά εμείς πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Ότι αλλιώ θα απορρίψουμε ολόκληρη την ε, πρόταση στο τέλος. Τέλο πάντων, ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα δείξει κοινή λογική στο μεταξύ. Αλλά σας το λέω. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί πάνω σε αυτό το σημείο. Πρέπει όλοι να στηρίξουμε τον εισηγητή και να ξέρουμε ότι κι εσείς είσαστε διατεθειμένοι αν φτάσουμε στο τέλος τη συνδιαλλαγή να απορρίψουμε την πρόταση εφόσον αυτό το σημείο δεν έχει γίνει δεκτό. Εύρος εφαρμογή τώρα. Εγώ δεν καταλαβαίνω εκατομμύρια και ένα αεροδρόμια να είναι πιο ασφαλή από άλλα αεροδρόμια που έχουν 4 εκατομμύρια 999.000 κλπ. επιβάτες. Εδώ δεν είναι θέμα νούμερων, είναι θέμα ασφάλειας. Δεν μπορεί να λέτε είναι θέμα ασφάλειας, γι' αυτό οι επιβάτες πρέπει να πληρώνουν και από την άλλη μεριά να λέτε πρέπει να βάλουμε κάποιο όριο γιατί ξαρτάται από τα νούμερα. Όχι. Αυτά συνδυάζονται. Τα κράτη-μέλη πληρώνουν. Δεν χρειάζεται όριο. Τα κράτη-μέλη πληρώνουν. Τελεία. Και εγώ στηρίζω αυτό που είπε και ο συγητής, αλλά και, και η κυρία Φώστερ, ότι όλα τα εμπορικά αεροδρόμια πρέπει να συμμετέχουν γιατί αλλιώς υπάρχει ένας αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα ασφάλειας. Κάθε εμπορική δραστηριότητα πρέπει να συμμετέχει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά με 5 εκατομμύρια να βάλουμε σαν όριο για μένα είναι μια ανόητη ιδέα, αγελία, όταν μιλάμε για ασφάλεια. Και ουσιαστικά είναι σαν να κρυβόμαστε επί στο δάχτυλό μας και να λέμε ναι, επειδή τα κράτη-μέλη δεν θα πληρώσουν, γι' αυτό λέμε να πληρώσει ο κόσμος. Όχι. Το θέμα είναι το ποιο πληρώνει. Αυτό πρέπει να δούμε. Γιατί άμα το αποφασίσουμε αυτό δεν έχει σημασία το όριο. Τα κράτη-μέλη θα πληρώνουν, οπότε όλα τα αεροδρόμια πρέπει να καλύπτονται. Σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Ο εισηγητή έχει κάνει πολύ καλή δουλειά για ένα τόσο δύσκολο και λεπτό θέμα. Πάντως, όπως είπαν και άλλοι, το έχουμε ξαναδεί αυτό και η κυρία Φώστερ και εγώ. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Όταν πήγε τελευταία φορά σε συνδιαλλαγή το κοινοβούλιο και παρετήθηκε, υποχώρησε. Όχι, αυτό να μην το κάνουμε αυτή τη φορά. Να μην υποχωρήσουμε. Και στο τέλος, αν το Συμβούλιο δεν δεχτεί το ποιος πληρώνει, τότε να απορρίψουμε ολόκληρη την πρόταση. Εντάξει, Εκ μέρους τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, κύριο Σίμπον, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και όλες. Επειδή είναι αυστριακός ο εισηγητής, μπορώ να χρησιμοποιήσω την γερμανική μητρική μου γλώσσα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Λάιχτφριντ, Έχουμε συζητήσει ήδη δύο φορέ το θέμα αυτό στην Επιτροπή Μεταφορών και μπορούμε να διαπιστώσουμε ήδη ότι οι στόχοι που επιδιώκει η Κομισιόν με την ρύθμιση αυτή του συμμερίζεται και η Επιτροπή σας, γιατί μόνο μέσα από μια οδηγία μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, να μην υπάρχουν αποκλίνουσες πρακτικές, να υπάρχει μια καλύτερη διαβούλευση με τους χρήστες των αεροδρομίων και να εξασφαλίσουμε ότι τα τέλη τα οποία θα επιβληθούν αντανακλούν το πραγματικό κόστος. Όλα αυτά είναι λοιπόν πολύ σημαντικά για την Κομισιόν. Θα ήθελα τώρα πρωτού διεξέλθω λεπτομεριακά σημεία να κάνω μερικές ε, γενικές παρατηρήσεις. Καταρχήν ο τομέας εφαρμογής. Αναφέρθηκε το θέμα αυτό από πολλούς ομιλητές. Το ζήτημα αυτό <clears throat> στη συζήτηση στο Συμβούλιο Υπουργών έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα γιατί η πλειοψηφία των κρατών μελών θα προτιμούσε να υπάρχει το κατόφλι των 5 εκατομμυρίων επιβατών και τώρα αυτό οδηγεί σε κάποιες ε, δυσκολίες για το γεγονός ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι το όριο αυτό του 5, των 5 εκατομμυρίων είναι πολύ υψηλό. <clears throat> και επίση το κείμενο για τα τέλη υπάρχει ένας περιορισμός γιατί όπως έχει ήδη αποφασιστεί από το δικαστήριο σε μια περίπτωση αγωγής, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα αεροδρόμιο σε κάθε χώρα το οποίο καλύπτεται. Οι νομομαθείς είπαν ότι δεν αποκλείεται να ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την άποψη ότι ένα κατόφλι μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις. Βάσει των στατιστικών, το όριο του 5, των 5 εκατομμυρίων σημαίνει ότι σε 7 κράτη-μέλη δεν θα εφαρμοστεί καθόλου αυτή η οδηγία. Κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό από την Κομισιόν. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι η πρόταση αυτής της Κομισιόν θα πρέπει να καλύπτει όλους, όλους τους εμπορικούς αερολιμένες. Τώρα, μπορεί παρόλα αυτά να υπάρξει ένα ενδιάμεσο όριο. Υπάρχει αυτή η πρόταση του ενός εκατομμυρίου επιβατών. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά κύριε Πρόεδρε, κύριε Λάιθριτ, νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι αποδεκτό από την Κομισιόν. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι το δύσκολο θέμα των διαφορετικών συστημάτων που ακολουθούνται στα κράτη-μέλη. Και αυτό έχει αναδυθεί στη συζήτηση έχουμε διαπιστώσει σε πολλά κράτη-μέλη όπου θα υπάρξουν αυτά τα τέλη, τα τέλη αυτά αποφασίζονται από τα ίδια τα αεροδρομία. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει απόφαση σε επίπεδο κυβερνήσεως ή σε περίπτωση κοινοβουλίου και αναφέρθηκε το, το παράδειγμα της Γαλλίας και της Ισπανίας, ακόμα και η Γερμανία έχει ένα σύστημα το οποίο προσωμιάζει με το γαλλικό και το ισπανικό. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν στην Κομισιόν να λάβει υπόψη όλα αυτά τα συστήματα στην πρότασή της και εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ανεξάρτητα από το σύστημα το οποίο ακολουθείται σε εθνικό επίπεδο να μην υπάρχει <clears throat> διάκριση αρνητική και να επιδιώκονται οι ίδιοι στόχοι σε όλα τα κράτη-μέλη. και γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι η αρμόδια επί της ουσίας υποστηρίζει ιδιαίτερα να υπάρχει η υποχρέωση στα κράτη-μέλη να χρηματοδοτούν όποια μέτρα ξεπερνούν τις ε, προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα χρηματοδοτούν από τους κρατικούς τους προϋπολογισμούς. Και έχετε διαπιστώσει Κύριε Πρόεδρε, αυτό που είπα προηγουμένω ότι είναι πολύ δύσκολη η συζήτηση που έχουμε με το Συμβούλιο των Υπουργών. Είναι σωστή η ανάλυση σα, αλλά εδώ πρέπει να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονό ότι δεν είμαι σίγουρο ότι ο κίνδυνο ο οποίο υπάρχει είναι να μην μπορούμε να επιτύχουμε την απαραίτητη διαφάνεια, την απαραίτητη έλλειψη ε, διακρίσεων. Το γνωρίζω αυτό. Αλλά εάν δεν γίνει δεκτή αυτή η πρόταση, αυτό το νομοθέτημα, τελικά τίποτα από όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε, διαφάνεια και ε, έλλειψη διακρίσεων, όλα αυτά θα εκπέσουν από μόνα του. Λοιπόν, θέλω να εκφράσω αυτό και να πω ότι είμαι ικανοποιημένο και με τη συζήτηση. Κύριε, ε, θα ήθελα να πω στον εκπρόσωπο τη Κομισιόν ότι αυτό που λέτε εγώ το περιμένω να το ακούσω από εσά για τα νέα μέλη της Επιτροπής. Κλασικό παράδειγμα τι γίνεται όταν πλησιάζουμε τη συνδιαλλαγή. Θα πούν μα θα σας δώσουμε αυτό, θα, θα σας δώσουμε εκείνο, μα θέλετε να απορρίψετε αυτό το νομοθέτημα και τι θα γίνει με τους φτωχούς επιβάτες. Την προηγούμενη φορά μας κοροϊδέψανε, την πατήσαμε, την φάγαμε. Ελπίζω να μην ξαναγίνει αυτό και πάλι. Κύριε Λάχτρου, έχετε το, το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα είμαι κάπως σύντομος. Θέλω ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις ε, συμβολές τους στη συζήτηση που θεωρώ ότι ήταν όλες επικοδομητικές. Σίγουρα θα πρέπει να οδηγηθούμε σε κάποια συμβαστική λύση σε ό,τι αφορά την ε, πληροφορία που δίνεται στους επιβάτες και τη συμμετοχή των επιβατών. Εμένα μου άρεσε ιδιαίτερα αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κούν γιατί και εγώ έψαξα να δω τι γίνεται σε σχέση με το κόστος και βρήκαμε μια πολύ ευρία ψαλίδα κόστους ε, επί τη βάση του ποια αεροπορική γραμμή εξετάζουμε από 1 ως 3 ευρώ κτλ. για το τι θα προκύψει ως πρόσθετο κόστος. Χαίρομαι επίσης και για το γεγονός ότι η Κομισιόν είπε σε σχέση με τον τομέα εφαρμογής, κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι απόλυτα λογικό. Δεν μπορούμε να έχουμε μια οδηγία που δεν εφαρμόζεται σε 7 κράτη-μέλη στην Ευρώπη. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει να το πούμε αυτό λοιπόν τελείως ανοιχτά. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε το γεγονός ότι τα εθνικά συστήματα έχουν τους λόγους τους να είναι διαφοροποιημένα. Εάν έχουμε την διαφάνεια, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί πρόβλημα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι ο στόχο τη διαφάνεια που θα πρέπει να έχουμε. Για την τροπολογία τώρα 29 και πάλι. Εγώ υποστηρίζω αυτό που είπε και ο πρόεδρός μας. Αλλά θέλω να προσθέσω και μία ακόμα σκέψη εδώ. Εμείς συζητούμε αφενός μία οδηγία η οποία αφορά το κόστος, το πρόσθετο κόστος για τα μέτρα ασφαλείας. Παράλληλα όμως, είναι δεδομένο ότι στους επόμενους μήνες θα υπάρξουν προτάσεις της Κομισιόν οι οποίες θα διατυπωθούν οι οποίες αφορούν απόλυτα τον τομέα εφαρμογής αυτών των μέτρων είναι οι σαρωτές σώματος, οι σαρωτές υγρών και τα λοιπά στα αεροδρόμια. Εγώ σας το λέω ειλικρινά. Δεν μπορούμε από τη μία πλευρά να προχωρούν τα πράγματα με τρομερή ταχύτητα και το Συμβούλιο να δείχνει μία διαθεσιμότητα να προχωρήσει με μεγάλη ταχύτητα, ενώ συγχρόνως θέματα χρηματοδότησης να μπλοκάρονται στο Συμβούλιο. Με την ψηφοφορία για το SWIFT Νομίζω ότι ακόμα και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει διαπιστώσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ίσες εξουσίες στον τομέα της νομοθεσίας και δεν είναι ένα σώμα το οποίο είναι δευτεροκλασσάτο. Γι' αυτό το λόγο εγώ θα ήθελα να προτείνω η Επιτροπή μας να ε, συζητήσει τι θα πρέπει να κάνει αν το Συμβούλιο δεν δείξει καμία θέληση να αντιμετωπίσει τα θέματα χρηματοδότησης αυτών των μέτρων. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο έχει νόημα τις οδηγίες αυτές που αφορούν την ασφάλεια στα αεροδρόμια, να τις συνδέσουμε με αυτή την οδηγία που αφορά το ποιο επομίζεται το κόστος της ασφάλειας στα αεροδρόμια. Αν δεν κινηθεί το Συμβούλιο λοιπόν να μην κινηθούμε ούτε και εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λέτφριτ. Πολύ διπλωματικό αυτό. Ναι. 1η Μαρτίου ψηφίζουμε στην Επιτροπή μας και τον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Επόμενο θέμα είναι η εφαρμογή του πρώτου πακέτου σιδηροδρόμων. Θα θυμόσαστε ότι η συζήτηση αυτή γίνεται μετά από συζήτηση που είχαμε τον Ιανουάριο οι συντονιστέ για να ζητήσουμε από την Επιτροπή να έχουμε μια συζήτηση για την εφαρμογή του πρώτου πακέτου σιδηροδρόμων. Το Δεκέμβριο είχαμε από την Επιτροπή τη δεύτερη έκθεση όσον αφορά την εποπτεία της ανάπτυξης της αγοράς. Πριν ζητήσω από την Επιτροπή να πάρει το λόγο, ξέρω ότι αυτό προέκυψε γιατί ακούγεται ότι η Επιτροπή μας, το Κοινοβούλιο, είναι δυσαρεστημένο για το επίπεδο εφαρμογής του πακέτου σιδηροδρόμων. Το ότι έχουν κάνει δηλαδή τα κράτη-μέλη μέχρι τώρα. Και γι' αυτό και ζητήσαμε να γίνει η συζήτηση αυτή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ακούσουμε από την Επιτροπή τι σκοπεύει να κάνει έτσι ώστε όλες οι χώρες μέλη να συμμορφώνονται προς τον νόμο, προς ό,τι έχει αποφασιστεί βάσει των διαδικασιών μας. Ο κύριος Πασχολή είναι εδώ, Βασκαρέλη. Ωραία. Ξέρω ότι δεν είναι τόσο ωραία όλα αυτά, αλλά πραγματικά πείτε μας τι θα κάνετε με τα κράτη-μέλη που δεν θέτουν σε εφαρμογή τις διατάξεις του πακέτου σιδηροδρόμων. Για να απαντήσω σύντομα, θα σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει διάφορες διαδικασίες επί παραβάση εναντίον των χωρών αυτών. Αυτή είναι η σύντομη απάντηση. Τώρα η πιο ε, μακριά απάντηση που έχω να σας δώσω είναι η εξής. Ακόμα και αν δεν έχει άμεση σχέση με αυτό που συζητάμε, πρέπει να ξέρετε ότι η Επιτροπή θέλει να εκφράσει τη θλίψη της για το τραγικό σιδηροδρομικό ατύχημα που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο Βέλγιο και όπου έχασαν τη ζωή τους 18 άνθρωποι. Τώρα, όσον αφορά την εφαρμογή του πρώτου πακέτου σιδηροδρόμων, όπως τροποποιήθηκε μετά από το δεύτερο και από το τρίτο, ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει τις εξελίξεις στην αγορά σιδηροδρόμων μέσω ενός μηχανισμού που ονομάζεται Rail Market Monitoring Scheme. Είναι ένα πρόγραμμα εποπτείας δηλαδή και η τελευταία σχετική έκθεση ε, ήταν έτοιμη το Δεκέμβριο του 2009. Από την έκθεση αυτή φαίνεται ότι υπάρχει μια θετική εξέλιξη στην αγορά αυτή για την περίοδο 2000 με 2009 που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του τελευταίου κομματιού 2000 από το 1990 μέχρι το 2000 και έχει να κάνει με τους επιβάτες, με τις υπηρεσίες προς τους ε, επιβάτες. Βέβαια υπάρχουν διαφορές ανάλογα με την περιοχή και μεγάλες μάλιστα πολλές φορές, ιδιαίτερα με τις χώρες εκείνες οι οποίες μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Οι προοπτικές εξέλιξεις της αγοράς σιδηροδρόμων είναι θετικές. Οι μελέτες μας δείχνουν ότι όντως όλο και μεγαλύτερο ρόλο παίζουν οι σιδηρόδρομοι, ότι συμπεριλαμβάνονται καλύτερα στις συνδυασμένε μεταφορές και ότι η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 έχει επηρεάσει σοβαρά, πολύ σοβαρά όλες τις μεταφορές, οπότε και τους σιδηροδρόμους. Και τόνισε ήδη υπαρχόμενα προβλήματα. Τώρα ποια είναι αυτά, ποιες είναι οι αδυναμίες των σιδηροδρόμων. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι το πρόβλημα είναι η αρχιτεκτονική χρηματοδότησης. Με τις οδηγίες μας, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να ισορροπούν τον προϋπολογισμό για τις υποδομές, που συχνά είναι μονοπόλιο, δεν ήταν πάντα. Ανήκουν πάντως οι υποδομές ως επιτοπλίστων στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη πρέπει να φροντίζουν να υπάρχει ισολογισμός στη διαχείριση. Ό,τι δηλαδή ε, δεν ε, φτάνει για τις υποδομές πρέπει να καλύπτεται από τα κράτη-μέλη. Να υπάρχει μια καλή τάξη και καλές υπηρεσίες προς όλους τους ενδυνάμει χρήστες. Δυστυχώς όμως αυτό δεν συμβαίνει παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι σιδηρόδρομοι. Δεν υπάρχουν αρκετές επενδύσεις όσον αφορά τις υποδομές. Πολλές χώρες μέλη επίσης δεν μπόρεσαν να αναπτύξουν σχέδια και να προγραμματίσουν την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων τους και έτσι δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αναδιάρθρωσης τόσο της διαχείρισης όσο και των υποδομών. Έπειτα, οι κανόνες όσον αφορά τις υποδομές διαφέρουν από χώρα σε χώρα κατά πολύ. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα έλεγα ότι είναι αρκετά ευρεία, δηλαδή επιτρέπει διακριτική μεταχείριση από τα κράτη-μέλη. Εμείς προσπαθούμε να βοηθούμε τα κράτη-μέλη να ερμηνεύσουν τους κανόνες και να τους εφαρμόσουν σωστά. Τέλος, συχνά, όχι πάντα, αλλά συχνά, οι υποχρώσεις των κρατών μελών ιδιαίτερα για τις μεταφορές στην περιφέρεια δεν ε, τηρούνται ε, σωστά. Δεν γίνονται έγκαιρα οι διαγωνισμοί, οι προκηρύξεις κλπ. Αυτά όσον αφορά την δημοσιονομική αρχιτεκτονική. Τώρα, άλλα στοιχεία αντικειμενικά που έχουν να κάνουν με τις αδυναμίες των σιδηροδρόμων. Τι φραγμοί υπάρχουν, τι δυσκολίες τεχνικής και οικονομικής φύσης υπάρχουν. Είναι ε, οι σιδηρόδρομοι ένα εντατικό οικονομικό εγχείρημα μπορώ να πω. Είναι κάτι που το βλέπουν όλοι, ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Και αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει επαρκής ρύθμιση. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάζουν βέβαια κανόνες αρκετά ξεκάθαρους, αλλά εφαρμόζονται διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Και μάλιστα τα ρυθμιστικά όργανα, που φυσικά έχουν διαφορετικές ονομασίες στις διάφορες χώρες, και παρακολουθούν την εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων δεν έχουν αρκετή εξουσία ή αρκετή ανεξαρτησία για να μπορούν να φέρουν σε πέρα στο έργο τους ικανοποιητικά ώστε να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες τελικά παντού σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Κάτι το οποίο δυσκολεύει τις, τον ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο. Το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια γενική έκθεση για την εφαρμογή του πρώτου πακέτου σιδηροδρόμων που ήταν μια περιγραφή της όλης κατάστασης. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν ε, έφτανε για να ξέρουμε τι γίνεται στις 25 χώρες μέλη τότε. Θελήσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Και έτσι προχωρήσαμε σε μια πολύ λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης στα διάφορα κράτη-μέλη με ερωτηματολόγια. Είχαμε καλή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και έτσι στη συνέχεια αποφασίσαμε να ε, εντοπίσουμε πιο συγκεκριμένα τις αδυναμίες των σιδηροδρόμων στην ευρωπαϊκή αγορά. Ξεκινήσαμε διαδικασίες επί παραβάση εφόσον είμαστε θεματοφύλακα των συνθηκών, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φροντίσει οι νόμοι να τηρούνται και να τίθεται σε εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Αυτός λοιπόν ήταν ένας τρόπος για να διορθωθούν μερικά στραβά στο σύστημα σιδηροδρόμων. Μετά αποφασίσαμε ότι έπρεπε να δούμε και την νομοθεσία ως έχει και να δούμε τι βελτιώσεις μπορούμε να επιφέρουμε. Ωραία διαδικασία επιπαραβάση λοιπόν για να διορθωθούν τα στραβά και μετά να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το πρώτο πακέτο σιδηροδρόμων. Όσον αφορά την διαδικασία επιπαραβάση, ξεκινήσαμε τον Ιούνιο του 2008 κατά 24 από τις 25 χώρες μέλη που έχουν σιδηροδρόμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι ένδειξη για το ότι είναι κακή η νομοθεσία μας. Επειδή κανείς δεν την τηρεί. Η νομοθεσία, έτσι όπως έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, υπάρχει και πρέπει να τηρείται. Η παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από τα κράτη-μέλη ήταν ε, διαφορετικού είδους, σε διαφορετικό βαθμό. Η κατάσταση δεν είναι άσπρο-μαύρο. Έτσι λοιπόν, στείλαμε και αιτιολογισμένες ε, συστάσεις το 2009 σε 21 από τις 24 χώρες. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι σε μία περίοδο ενός έτους, ουσιαστικά, είχαμε έναν πολύ εντατικό διάλογο με όλες τις χώρες μέλη. Στόχος μας με τη διαδικασία επιβαραβάσης δεν ήταν να πάμε τις χώρες στο δικαστήριο, αλλά να φροντίσουμε ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία ορθά. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και είχαμε συναντήσεις μαζί τους όπου συζητήσαμε βελτιώσεις ή αλλαγές στην νομοθεσία ή στην πρακτική ορισμένων χωρών. Και πετύχαμε κάποια αποτελέσματα. Όχι μόνο τρεις χώρες ε, μέλη ξέφυγαν από το δεύτερο στάδιο της ε, αιτιολογημένης γνώμης, αλλά επιπλέον περιορίσαμε το εύρος των ε, διαδικασιών επί παραβάση και στο μεταξύ ορισμένες χώρες έβαλαν κάποια τάξη στη κατάσταση. Τώρα, τι θέλαμε να διορθώσουμε με τις διαδικασίες επί παραβάση. Πρώτα απ' όλα το θέμα των ε, υποδομών. Υπάρχει νομοθεσία η οποία δέχεται να μην είναι κανείς τέλειος όταν πρόκειται για τον υπολογισμό των τελών υποδομών. Ε, οι αρχές πρέπει να βάζουν κανόνες και να υπολογίζουν τα τέλη υποδομών. Αυτός λοιπόν είναι ένας τομέας όπου υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία μεταξύ των κρατών μελών. Ο βασικός κανόνας είναι ότι τα βασικά τέλη υποδομών πρέπει να είναι το... η διαφορά ανάμεσα στο κόστος που προκύπτει από το δίκτυο, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να το υπολογίσουμε ακριβώς αυτό το περιθώριο. Πρέπει να βρούμε λοιπόν κριτήρια και έπειτα επιτρέπονται κάποιες διαφορές όσο τις αντέχει η αγορά. Όσο δεν υπάρχει κομμάτι των σιδηροδρόμων που να αποκλείεται από τις υποδομές. Τα κράτη-μέλη και όσοι ασχολούνται με αυτό δεν ε, το δοκιμάζουν αυτό. Δεν ξέρουν αν το αντέχει η αγορά ή όχι. Και εκεί μερικές φορές έπρεπε να τους επαναφέρουμε στην τάξη. για το κατά πόσο είναι αποδεκτά ή όχι τα τέλη υποδομών. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες για προγράμματα απόδοσης, για το πώς μοιράζεται η ευθύνη στις καθυστερήσεις που γίνονται και πώς αντισταθμίζεται η άλλη πλευρά η οποία δεν είναι υπεύθυνη για τις καθυστερήσεις ή για, τις, για τη ζημιά. Ένας δεύτερος τομέας που μας απασχόλησε ήταν η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομών. Είναι ανεξαρτησία δηλαδή της αρχής της υπεύθυνη για τις κύριες λειτουργίες. Που ποιες είναι? Είναι οι διαδρομές και τα τέλη για τη χρήση των υποδομών. Σε μια ανοιχτή αγορά, σε μια αγορά που βρίσκεται σε ανταγωνισμό, αυτές οι βασικές λειτουργίες δεν είναι δυνατόν να ασκούνται από μία αρχή, από μία οντότητα, η οποία να συνδέεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με ε, την επιχείρηση σιδηροδρόμων. Γιατί τότε καταλαβαίνετε ότι αυτός που πληρώνει και αυτός που πληρώνει συνδέονται. Δεν μπορούμε αυτό να το δεχτούμε. Γι' αυτό και υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την ανεξαρτησία των βασικών λειτουργιών με πολύ σαφείς όρους. Κάτι όμως το οποίο δεν τηρείται επαρκώς από τα κράτη-μέλη. Εδώ δεν ε, είναι η κάθετη διάκριση στα holding ανάμεσα στη διαχείριση των υποδομών και την επιχείρηση σιδηροδρόμων, γιατί ακόμα και στη περίπτωση που υπάρχει πλήρης διάκριση υπάρχουν προβλήματα επειδή δεν υπάρχει ανεξαρτησία στην άσκηση των βασικών λειτουργιών. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την σωστή λειτουργία μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς. Έρχομαι τώρα στον τρίτο τομέα ανησυχίας μας, που έχει να κάνει με την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών οργάνων. Αυτός που ρυθμίζει το ισόπεδο του γηπέδου είτε δεν είναι αρκετά ανεξάρτητος, διότι αποτελεί τμήμα του συστήματος μέσα στο οποίο είναι εμβαπτισμένος, δηλαδή του συστήματος που εξασφαλίζει τη λειτουργία των σιδηροδρόμων, είτε σε άλλες περιπτώσεις δεν έχει τους απαραίτητους πόρους για να εφαρμόσει την ρυθμιστική αυτή λειτουργία ανθρώπινου ή υλικού πόρου ή και του δύο. Και εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν τι απαραίτητε ικανότητε. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναθεώρηση, δηλαδή τι δραστηριότητε που έχουμε ξεκινήσει για να βελτιώσουμε την ποιότητα τη νομοθεσία, Καταρχήν έχει τροποποιηθεί το πρώτο πακέτο σιδηροδρόμων, το δεύτερο έχει επίση τροποποιηθεί από το τρίτο πακέτο σιδηροδρόμων. Είναι σιδηρόδρομο η ίδια η νομοθεσία. Είναι δύσκολο να την αναγνώσει κανεί, Είναι κατακαιρματισμένη σε διάφορα νομοθετήματα. Υπάρχουν πολλοί κανόνε οι οποίοι αφορούσαν μεταβατικέ περιόδου. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο κώδικα για του σιδηροδρόμου. Θα πρέπει σε ένα ενιαίο κείμενο να ενσωματωθούν 5, 6, άντε και 7 ίσω οδηγίε για να γίνουν αναγνωσιμότερε και προσβασιμότερε. Θέλουμε συγχρόνως να αποφύγουμε δογματικού χαρακτήρα συζητήσεις οι οποίες μπορεί να γοητεύουν και να μαγεύουν τους σιδηροδρομάδες σε όλη την Ευρώπη, αλλά εμείς θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων σε πέντε ή έξι πρωτοβουλίες που για μας είναι σημαντικές για να εξασφαλίσουμε την ισότητα ανταγωνισμού. Τα θέματα χρηματοδότησης, τα θέματα τιμολόγησης, η τιμολόγηση για τη χρήση των υποδομών δηλαδή, η πρόσβαση στις υπηρεσίες, όχι τόσο στην ικανότητα των σιδηροδρόμων ή στην υποδομή των ε, σιδηροδρόμων, των υποδομών, το τελευταίο μηλι η πρόσβαση στα, στους σιδηροδρομικούς κόμβους στον ε, διαχειριστή υποδομών ο οποίος δεν είναι απόλυτα ανεξάρτητος από τους ε, φορείς λειτουργίας των συνδεδόμων. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον νεόφερτο να έχει πρόσβαση σε ουσιαστικές υπηρεσίες για να λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία, να μπορούν να μετακινούνται από γραμμή σε γραμμή τα βαγόνια, παραγματικά χάρη στους σταθμούς μετα... μετακίνησης, να αναφοδιάζονται οι σιδηροδρόμοι με καύσιμο. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε και την ικανότητα των ρυθμιστικών αρχών να δρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κόντευω να τελειώσω κιόλα. Λοιπόν, πότε θα τα προτείνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Θα ζητήσω αύριο το απόγευμα από τον Επίτροπο Κάλλα να μα πει. Δεν έχει ακόμα αποφασιστεί για τις υπηρεσίες. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Δεν θέλουμε να παραφορτώσουμε τη βάρκα με πάρα πολλά θέματα τα οποία θα είναι επίμαχα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα ουσιαστικά για να λειτουργήσει καλύτερα η αγορά. Και εν παραλίλω έχουμε μια ολιστική αντιμετώπιση στους σιδηροδρόμους. Το πρώτο πακέτο καλύπτει τις οικονομικές πτυχές, αλλά συζητούμε επίσης και για την διαλειτουργικότητα, την κοινή αποδοχή, για την ε, αποτροπή των ατυχημάτων όπως αυτό του Χάλε, παρόλα αυτά παραμένουν σιδηρόδρομοι πολύ ασφαλέστεροι από τις οδικές μεταφορές. Μπορούμε να κάνουμε πολλά για να γίνουν ακόμα ασφαλέστεροι, αλλά προσπαθούμε να αναζωογονήσουμε τη χρήση των σιδηροδρόμων για εμπορευματικές μεταφορές κατά, την, κατά μήκος των διαδρόμων και είναι σε δεύτερη ανάγνωση ενώπιον του Κοινοβουλίου αυτό το θέμα. Πάντα με εκπλήτη το ότι στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα εργαζόμαστε ακόμα με κανόνες οι οποίοι ανατρέχουν στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Εξακολουθώ να ελπίζω πάντως παρόλα αυτά. Κύριε Γκρός, πάρα πολλά θα μπορούσα να πω κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο όμως. Το ξέρω, το ξέρω ότι και εσείς αυτό θέλετε. Θα έλεγα ότι διαβάζοντας αυτή την έκθεση της Κομισιόν έχω την εντύπωση ότι οι σιδηρόδρομοι είναι αρμοδιότητα των Υπουργείων Άμυνα πολλών κρατών μελών και όχι του Υπουργείου Μεταφορών. Γίνονται τόσο μεγάλες προσπάθειες σε κάθε χώρα να διαφυλάξουν ως κόριο οφθαλμού την αυτονομία των ε, σιδηροδρόμων. Και φαίνεται ότι ο φορέας ο οποίος παρέχει υπηρεσίες είναι πιο σημαντικός από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. Αυτό το οποίο είναι ουσιαστικό είναι ότι όταν τα κράτη-μέλη δέχονται μία νομοθεσία θα πρέπει να συμβάλλουν στο να υπάρξει και μία ευρωπαϊκή πολιτική η οποία είναι αξιόπιστη. Δεν Μπορούμε όμως να προχωρήσουμε όταν το Συμβούλιο κάνει τόσο μεγάλες προσπάθειες να μην εφαρμόσει αυτά τα οποία συμφωνεί. Πιστεύω ότι από την πλευρά του Κοινοβουλίου θα πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν νέα μέσα και νέες προσπάθειες για να προχωρήσουν όλα αυτά που είναι στα συνδρομικά πακέτα γιατί είναι θέμα αξιοπιστίας για την παραβίαση των συμβάσεων, για το θέμα των τελών. Ο κύριος Κράμετα έχει αναφέρει αυτά τόσες πολλές φορές, το θέμα της ανεξαρτησίας, η πολυπλοκότητα των δομών των συνδρομικών επιχειρήσεων. Και το ερώτημα το οποίο εγώ θα ήθελα να θέσω, η φιλελευθερωποίηση οδήγησε σε αποτελεσματικότητα, διαλειτουργικότητα ή ασφάλεια. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά ξεδιάντροπο εμείς θα έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την ε, νομοθεσία και την εφαρμογή της στα κράτη-μέλη και στην περίπτωση μη εφαρμογής της να λαμβάνεται αυτό υπόψη τουλάχιστον σε κάθε επίπεδο. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι παράλογο. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ακριβώς να εφαρμόζονται αυτά τα οποία αποφασίζουμε και στη συνέχεια να υπάρχει και μία σειρά προτεραιοτήτων. Δεν είναι μονάχα η αποτροπή των ατυχημάτων, αλλά και για μένα η διαλειτουργικότητα. Και θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τη σαφή απάντηση που μας έδωσαν. Που έδωσε για το ατύχημα, γιατί πολλές φορές οι επιχειρήσεις ψάχνουν κάποιο αποδιοπομπαίο τράγο όταν γίνεται ένα ατύχημα και θεωρούν ότι έτσι αποσύουν τις ευθύνες τους να εφαρμόζουν κοινά στάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε την διαλειτουργικότητα. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο βασικές άποψες και ελπίζω ότι αύριο με ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μπορούμε να μιλήσουμε όπου θα υπάρχει κοινή ευθύνη όλων των κρατών μελών. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν και η ελπίδα μου είναι ότι η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο θα μπορέσουν να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση και να μπορέσουν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τα υπεσχημένα και τις υποχρεώσεις που έχουν υπογράψει. Ξέρω ότι δεν ήσασταν παρόν εδώ κύριε Γκρός χθε, αλλά χθε που είχαμε ενός λεπτού σιγή για το ατύχημα είπαμε πολύ διπλωματικά ότι μας απογοήτευσε η στάση του Βελγίου σε σχέση με το ατύχημα και τις ευθύνε. Γιατί πολλοί θεώρησαν ότι έπρεπε να καταλογίσουν ευθύνε προτού ακόμα εκδοθεί η επίσημη έκθεση. Κύριε Αλ Καντράουι και άλλα τρία άτομα. Έχουμε εννέα λεπτά παρακαλώ να είσαστε πολύ σύντομοι. Όλοι θέλετε να πείτε κάτι, αλλά ούτως ή άλλως θα συζητηθεί το προφορικό ερώτημα που σχετίζεται με τα θέματα αυτά και θα έχετε περιπλέον χρόνο για συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά βέβαια θα μπορούσα να πω, θα περιοριστώ όμως σε κάποια μόνο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα για την αξιολόγηση. Δύο τρόπους μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ή να δούμε τι γίνεται με την νομοθεσία, πώς έχει εξελιχθεί, ή μπορούμε να δούμε τους στόχους μας. Τους έχουμε πετύχει. Επ' αυτού λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά τους σιδηροδρόμους, και τις εμπορικές μεταφορές. Υπάρξει κάποια σταθεροποίηση τα τελευταία χρόνια, δεν έχω βέβαια και τα εντελώ πρόσφατα στοιχεία. Όσον αφορά όμως τους επιβάτες, εδώ υπάρχει μια μικρή άνοδος. Οπότε εγώ αναρωτιέμαι το άνοιγμα της αγοράς που εντάξει για τα εμπορεύματα βοήθησε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί σιδηρόδρομοι και αν όχι, τι φταίει. Πάντα έλεγα ότι ο ανταγωνισμός στους σιδηροδρόμους δεν έχει να κάνει μόνο με το άνοιγμα της αγοράς, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνδυαστεί και με τις ε, πολύτροπες μεταφορές. Ότι χρειάζεται ένας άλλος μηχανισμός για να μπορέσουν να πετύχουν οι συνδυασμένες μεταφορές. Το συμπέρασμά μου είναι ότι εφόσον θέλουμε να πάμε ακόμα πιο πέρα όσον αφορά τις μεταφορές επιβατών, πρέπει να καθίσουμε να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες, να δούμε οι δημόσιες υπηρεσίες τι προσφέρουν και να είμαστε έτοιμοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο να επικρίνουμε και το άνοιγμα της αγοράς ενδεχομένως εφόσον είναι σε βάρος κοινωνικών προδιαγραφών, εργαζομένων κλπ. Τέλος, Πρόεδρε, συμφωνώ ότι πρέπει να κοιτάξουμε στα κράτη-μέλη τι γίνεται και να φροντίσουμε να ενισχύσουν την υπηρεσία αυτή και να υπάρχει καλή ρυθμίση της αγοράς. Οι εθνικές αρχές όμως πρέπει να κοιτάνε και την ασφάλεια και τις συνδυασμένε μεταφορές. Είναι και αυτά πράγματα που πρέπει να έχουν υπόψη τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάμερ, δύο λεπτά παρακαλώ. Φυσικά ξέρουμε όλοι ότι είναι το τελευταίο εθνικό προπύργιο οι σιδηρόδρομοι που με νύχια και δόντια το προστατεύουν και δεν θέλουν να το αφήσουν να περάσει σε ευρωπαϊκές δομές. Αλλά κάτι πρέπει να είναι σαφές σε όλους. Είχαμε καταφέρει κάποια πράγματα. Ξέρουμε ότι η φιλελευθερωποίηση στον αεροπορικό τομέα έφερε τεράστια ανάπτυξη, περισσότερη από ό,τι θα ήθελα εγώ σαν ε, πράσινος. Στην περίπτωση της, ε, των σιδηροδρόμων, τα πράγματα είναι σαφή ότι με την φιλελευθερωποίηση των εμπορευματικών μεταφορών η Ολλανδία συν 40% ανέβηκε η κίνηση, συν 30% στην Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο 60%, 20% στη Γερμανία. Λοιπόν, όλα αυτά προχώρησαν. Ενώ η Γαλλία που έμεινε αποκλεισμένη από τις άλλες χώρες και τη φιλελευθερωποίηση μειώθηκε η κυκλοφορία κατά 28%. Και η Γαλλία τι πέτυχε έχασε θέσεις ε, απασχόλησης, μεταφέρθηκαν μεταφορές στον δρόμο γιατί θεώρησαν ότι το να μην φιλελευθερωποιήσουν θα ήταν καλύτερο. Δεν ήταν καλύτερο, ήταν χειρότερο. Πρέπει να λάβουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη μας και στη δημόσια συζήτηση το άνοιγμα των δικτύων οδηγεί σε μεγαλύτερη κυκλοφορία στους σιδηροδρόμους. Ελοχεύει βέβαια και ο κίνδυνος αν υπάρχει πάντα η κερδοφορία ως ύψιστος γνώμων ότι δεν κατέστρεψε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, το κατέστρεψε το S-Bahn στο Βερολίνο, γιατί το μόνο πράγμα που τους ένοιαζε ήταν να έχουν περισσότερο κέρδος. Λοιπόν, οδήγησε αυτό σε πάρα πολύ ακριβές αστικές συγκοινωνίες. Αφήνουν το κράτος να είναι υπεύθυνο για τις υποδομές και απλώς παίρνουν το κέρδος από τη λειτουργία της ε, τις λειτουργίες. Στο Βέλγιο όταν υπάρχει ένα κόκκινο φως το οποίο το περνάει, ένα κόκκινο φανάρι το οποίο το περνάει το τρένο, θα πρέπει να υπάρχει ο μηχανισμός ο οποίος το σταματάει αυτόματα. Αυτό η τεχνολογία υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Λοιπόν, στην Κομισιόν σας λέω, πρέπει να δράσετε. Έχετε δικαιώματα, είσαστε ο θεματοφύλακας των συνθηκών. Τι κάνετε όμως. κάνετε εκθέσεις που ουσιαστικά τις παραβιάζουν 24 από τα 25 κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει με τέτοιους τρόπους να γίνονται ε, μεταφορές οι οποίες παραβιάζουν τους κανόνες. Η Γαλλία κρατάει συγκεκριμένα σλότ για τον εαυτό της τα οποία δεν τα χρησιμοποιεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι μειώθηκε η δραστηριότητα. Λοιπόν αυτό είναι μια παραβίαση των κανόνων, μια κατάχρηση των κανόνων. Εσείς έχετε λοιπόν το, το καθήκον να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις για όλα αυτά τα θέματα. Και έχετε όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία σας έδωσα. Η κυρία Ντουράουν, τελευταία ομιλήτρια, αν μπορείτε να παραμείνετε σε πολύ, στα δύο λεφτά που μένουν, είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιες αποφρώσεις μονάχα. Νομίζω ότι όταν οι 24 χώρες ε, επί 25 βρίσκονται σε διαδικασία παραβάσεως, ε, αυτό κάτι σημαίνει. Παρατηρήσεις μου λοιπόν. Πρώτον, είτε ξεκινάμε από το γεγονός ότι η φιλελευθερωποίηση έγινε το η πρώτη δέσμη, δηλαδή έγινε, προχώρησε και δεν κατάφεραν οι χώρες να ρυθμίσουν τα θέματα καλά ε, και εν πάση περιπτώσει δεν θα έπρεπε να είχαμε δεχτεί ο επόπτης να είναι ε, μέσα στην επιχείρηση, να είναι εκτός επιχείρησης έτσι ώστε η ρύθμιση να γίνει από μια πραγματικά ανεξάρτητη αρχή. Πέραν τούτου όμως νομίζω ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα και πιστεύω ότι η αύξηση του αριθμού των ε, επιβατών έγινε χωρίς φιλελευθερωποίηση και όσον αφορά ε, την μεταφορά φορτίων θα πρέπει να δούμε. Ενδεχομένως στη Γερμανία να είχαμε ανάπτυξη αλλά σε άλλες χώρες όχι. Έχουμε μάλλον συγκέντρωση παρά ε, κατακαιρματισμό, δηλαδή παρά μεγαλύτερο ρυθμό μικρών νεοεισερχόμενων. Δηλαδή τι θέλουμε. Θέλουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση σιδηροδρόμων ή θέλουμε πληθώρα μικρών, ε, μικρών που θα εμπλουτίσουν τους σιδηρόδρομους. Εγώ νομίζω ότι πριν προχωρήσουμε περαιτέρω στην φιλελευθερωποίηση των επιβοτών που με βρίσκει κάθετα αντίθετη γιατί τίποτα δεν μπορεί να μας αποφύρει. Εάν ε, μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα ακόμα αυτό όσον αφορά τη μεταφορά φορτίων, οπωσδήποτε είμαι αντίθετη όσον αφορά την μεταφορά επιβατών. Πιστεύω ότι αυτά τα τρία επόμενα πακέτα θα πρέπει εκβάθρον να θεωρηθούν έτσι ώστε να μην έχουμε τις ίδιε καταστροφικές συνέπειες στις δημόσιες υπηρεσίες. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. ε, ε λοιπόν, όπως σας είπα, σας ζήτησα να είστε σύντομοι, θα έχουμε μια προφορική ερώτηση όσον αφορά ε, το θέμα αυτό και μπορούν άνετα να εκδηλώσουν το άγχος τους και τον προβληματισμό τους στα μέλη ε, σε, ε, στα πλαίσια αυτής της συζήτησης, της προφορικής ερώτησης, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο υποβόσκον άγχος, βλέπε αγανάκτηση στην Επιτροπή μας εδώ. Φαίνεται ότι πολλά πράγματα δεν γίνονται καλά, πολύ μεγάλη ε, μεγάλη αγωνία υπάρχει από πλευράς ε, των ε, κρατών που από τη μία πλευρά ψηφίζουν κάποιους κανονισμούς μετά όπως είπε και ο κύριος Κράμερ επανεθνικοποιούν έτσι ώστε να οπισθοδρομήσουν. Όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε εκτενώς στην προφορική ερώτηση. Πάντως σας ευχαριστούμε που ήρθατε και μας δώσατε την πληροφόρηση για το που βρίσκεται η συζήτηση. Λοιπόν, ε, κατανοώ ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έτσι μια, ένα άγχος όσον αφορά το ίδιο θέμα. Λοιπόν, επόμενη συνεδρίαση, Δευτέρα απόγευμα, 1η Μαρτίου στις 3 στις Βρυξέλλες. Θα έχουμε μονάχα εκείνο το απόγευμα συνεδρίαση. Ευχαριστούμε όλους, ευχαριστούμε και τους διερμηνείς και όλο το προσωπικό. Γεια σας.